we Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε αν θέλετε με λίγη ησυχία να παρακαλέσω. Καλώς ήλθατε όλοι τα μέλη της Επιτροπής, οι ελεγκτές. Ελπίζω να είχατε καλές θερινές διακοπές. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα πίσω στα Θρανία. Και συνεχίζω στα Ιταλικά, λέει τώρα η Πρόεδρος, στα Ιταλικά. Σήμερα έχουμε λοιπόν ένα απόγευμα αρκετά γεμάτο και πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε πολλά να αποφασίσουμε και για την συνάντηση των συντονιστών. Τώρα, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα θεωρήσω ότι έχει εγκριθεί το σχέδιο μισή διατάξεως. Δεύτερον, θα θεωρήσω, εφόσον δεν έχουμε σχόλια, και τα πρακτικά της 20 Ιουνίου εγκεκριμένα. Σήμερα έχουμε διερμηνία με σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Ευχαριστεί και τους Ελληνείς ευγενικά η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και εμείς. Έχουμε web streaming βεβαίως. Και να θυμίσω επίσης ότι τα πρακτικά της 13ης, 13ης ε, Ιουλίου έχουν ήδη εγκριθεί, δεν έχουμε άλλες ε, αντιρρήσεις, δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις μέχρι εντός της προθεσμίας μάλλον. Να ξεκινήσω τώρα από μια λεπτομέρεια που όμως είναι σημαντική για μένα. Ε, θα γνωρίζετε ότι μας έπληξε στη χώρα μου ένας ε, βιώτατος σεισμός με πολλά θύματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και των άλλων οργάνων όλους εκείνους που εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους. Να σας ενημερώσω επίσης ότι εγώ ήμουν, επισκέφτηκα τις ε, οικογένειες των θυμάτων και βεβαίως τη χώρα, η κυβέρνηση, οι τοπικές αρχές ε, όλοι ε, κάνουν κάθε προσπάθεια. Είμαι βέβαιη ότι και οι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δεσμικά όργανα θα εκφράσουν και εμπράκτο την υποστήριξή τους με την κινητοποίηση και των σχετικών μέσων και θα το πω και σε εσά ε, εντός μηνός, του ερχομένου μηνό, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία για να εξακριβώσουμε πώς πάνε τα πράγματα και ε, για, τους, για τα θύματα και τι οικογένειε του. Υπάρχει και ένα φόρουμ ε, που προωθεί η Κομισιόν για τα ακουστικά στην ε, Βενετία και είχαμε και εκπροσώπηση και νικητές από το Μπενελούξ. Αυτό θα έχουν την ευκαιρία τους τρεις ε, βραβευθέντες να τους δούμε όλοι, τις συμμετοχές αυτές. Πρόκειται για εξαιρετική δουλειά και οι 28 νεαροί σπουδαστές ε, συνεφίλ ε, στη Βενετία συμμετείχαν πολύ ενεργά και για το φόρουμ οπτικοακουστικών αυτό ήθελα να πω απλώς. Εγώ ήμουν εκεί μαζί με την αντιπροσία της Κομισιόν και ο κύριος Μόργανο και η κυρία Έλερ. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με δύο τίτλους για το νέο χρηματοδοτικό μέσο που προβλέπεται για τη Δημιουργική Ευρώπη. Έγινε εμβάθυνση και συζήτηση από αυτού. Ξέρετε ότι 30 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία του διαγωνισμού, μάλλον της υποβολής υποψηφιωτήτων για το ταμείο αυτό, για το μέσο αυτό. Εμείς ε, συμμετέχουμε και παρακολουθούμε ενεργά. Και ο άλλος τίτλος είναι ο διαφορετικός ρόλος ε, που μπορούν και πρέπει να έχουν οι κινηματογραφικές αίθουσες στην Ευρώπη ως ε, χώροι συνάθρησης αλλά και ενημέρωσης γενικώ. Επίσης, 8 Σεπτεμβρίου να πω, θα έχουμε ένα σεμινάριο Επιτροπής ε, Πολιτικών Θεμάτων και ΕΜΠΛ ε, για να συνεχίσουμε τη συνεργασία που έχουμε οι δύο επιτροπές και που την θέλαμε όλοι για το θεματολόγιο, για τις αρμοδιότητες, μάλλον για τις δεξιότητες, ε, με θεματικές ε, παρουσιάσεις. Το πρόγραμμα έχει ήδη κυκλοφορήσει. Ωστόσο, εγώ λόγω απροόπτου δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω και θα ευχαριστήσω ήδη την αναπληρώτη. Ε, Σβοϊντρόβα για την αντικατάσταση και θα ήθελα να πω ότι εμείς πρέπει να προσέξουμε και αυτό το θέμα και να συμμετάσχουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τώρα, να χαιρετήσω τον κύριο Φοντάνη και τους άλλους συναδέλφους της UNESCO. Θυμίζω την ε, Διεθνή ημέρα του, κατά του αναφαλβετισμού είναι μια πολύ σημαντική μάχη, πόλεμος αν θέλετε, που δεν έχουμε κερδίσει ακόμα. Η μέρα που διακηρύχθηκε ε, το 76. Είμαστε λοιπόν στην 50η επέτειο. Και φαίνεται απίστευτο, αλλά ακόμα έχουμε τέτοια σημαντικά κρούσματα. Διαβάζουμε το παρελθόν, γράφουμε το μέλλον, ε, λέγεται η σχετική εκστρατεία προώθησης μαζί με το υλικό που έχετε μπροστά σα σχετικά με αυτό. Μια σημαντική ευκαιρία για τη διεθνή κοινότητα λοιπόν να χαιρετήσει και τα μαθήματα και τις επιτυχίες που είχαμε αλλά να επανεκκινήσουμε στους στόχους επί των οποίων χρειαζόμαστε περισσότερο δουλειά. 75 εκατομμύρια ενηλίκων είναι αναλφάβητοι αυτή τη στιγμή, 17% δηλαδή του παγκόσμιου πληθυσμού των ενηλίκων. Δύο τρίτα εξ αυτών είναι νεαροί και γυναίκες. Επομένως έχει σχέση και με την Ευρώπη αυτό. 122 εκατομμύρια νεαροί σήμερα δεν μπορούν να γράψουν την πιο απλή φράση. Μεταξύ των οποίων και γυναίκες που σε πολλές χώρες είναι η πλειοψηφία των διπλωματούχων, αλλά εδώ είναι το 70%. 77 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο και επομένω κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ δύσκολο μέλλον και στην πολιτικοστή αυτή επέτειο μου φάνηκε σημαντικό να μην είμαστε αδιάφοροι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα και να βρούμε τους τρόπους για να συνεργαστούμε ακόμα καλύτερα και με την UNESCO και με τους άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία αυτή και να τονίσω ότι ο αλφαβητισμός είναι παγκόσμιο δικαίωμα για όλους. Τώρα, πάμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία για την ε, γνωμοδότηση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Στρογέσκη ε, για τη δουλειά. Αν έχετε την κάρτα, έχουμε την έγκριση του προϋπολογισμού 2017 τις τροπολογίε και το σχέδιο γνωμοδότηση έκθεση. δύο διαφορετικές πληροφορίε. άρα πάμε αμέσως στην ψηφοφορία. Ήθελα όμως να δω μήπως ο συνάδελφος θα ήθελε να πει δύο λόγια εισαγωγικά. Όχι, ε, εντάξει, πάμε ευθεία στην ψήφο λοιπόν. Είστε όλοι έτοιμοι λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από τις τροπολογίες. Ε, η επαριθμόν 63-50. Α, ποιος είναι υπέρ. 63-50 επαναλαμβάνω. Κώστα Μόργανο. Μιλάμε για τα draft budgetary amendments, λέει η Πρόεδρος. Όχι όχι τον άλλο κατάλογο, τις τροπολογίες. 63-50 λοιπόν. Η πρώτη. Κώστα και Μόργανο. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 63-52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63-93 υπέρ κατα εποχες αποχές εγκρίνεται. 63-94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-96 όχι. Α, όχι, ναι. Άρα πάμε στην 63-66. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63-55. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-59 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. I close Πέρασε. Εγκρίνεται. Όχι, όχι. Απορρίπτεται. Διορθώνει η Πρόεδρος. 14-12. Λοιπόν, 63-60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 63-61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 64-04 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνει 64-05 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64-06 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64-07 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64-12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64-08 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63-62 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63-63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63-64 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 63-67 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63-68 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αλλά ας το ελέγξουμε άρχιτη ψηφοφορία πέρασε ψηφοφορίες απορρίπτεται 63-69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63-70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6371 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6372 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αλλά να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία 6372 For me uh, I the vote. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, λέει η πρόεδρος. Α, όχι, όχι, απορρίπτεται. Λοιπόν, 63-73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτει. 63-74 υπέρ. Κατά αποχές 6375 υπέρ κατά αποχές 6376 υπέρ κατά αποχές 6377 υπέρ κατά αποχές 6379 υπέρ κατά αποχές 6380 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63, 81 υπέρ. Κατά, ξανά υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και επομένως πάμε στην 63-82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και επομένως πάμε στην 63-84 υπέρ. Κατά

4. 09 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64-10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64-11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 64-00 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64-15 από υπέρ κατα αποχή αποχές εγκρίνεται. Άρα 64-01 υπέρ αποχή αποχές εγκρίνεται. 64-16 υπέρ αποχή αποχές εγκρίνεται. 64-03 του εισηγητή υπέρ αποχή αποχές εγκρίνεται. 63-89 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Close the vote. Πέρασε. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 63-97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 63-90 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 63-91 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 63-92 η τελευταία. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Πάμε στο δεύτερο έγγραφο. Παράγραφος 1, τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τέσσερα υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία για την 4 πέρας εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έξι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 έχει ζητήσει το Λαϊκό Κόμμα split vote εδώ υπέρ κατά για το πρώτο κομμάτι έτσι εγκρίνεται δεύτερο το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δύο ε ή εννέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Για την 11, άρχεται. Για την 11 λέμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε θέλετε. Γιατί 14 λοιπόν ελέγχουμε. Παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για το σύνολο τώρα της, ε, του σχεδίου άρχεται η ψηφοφορία και πέρας της ψηφοφορίας ταυτόχρονα. 20 in favor, 20 υπέρ, 2 κατά και 2 εποχές συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστούμε συνάδελφε. για τη δουλειά αυτή τον κύριο Δρογεύσκη που έδωσε μάχη στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού. Continuiamo. Ε, colleghi. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα έχουμε... Ζητώ συγγνώμη ένα λεπτάκι να καλέσω την καλέσαμε έτσι δεν είναι ένα λεπτάκι γιατί εδώ οργανωνόμαστε για να έχουμε τους τρεις ερευνητές για την έρευνα για την εφαρμοστική έκθεση της Δημιουργικής Ευρώπης εγώ είχα κάνει μια εισαγωγή με συζήτηση στις 14 Ιουλίου την τελευταία φορά που συναντήκαμε. Oh, nice to meet you. Nice to, no, nice to meet you. Okay, the other ones, the others are coming. And so, Λοιπόν, όπως ξέρετε, έχουμε ήδη ξεκινήσει τη συζήτηση επί δύο εκθέσεων εφαρμογής 13 και 14 Ιουλίου για το Εράσμος με τα αποτελέσματα των ερευνών που είχαν τεθεί στο κατάλληλο τμήμα και την Δημιουργική Ευρώπη. Και υπήρξε και μια δυσκολία για να βρούμε όλους τους ερευνητές και ήταν η τελευταία συνάντηση με όχι σημαντική συμμετοχή των μελών. Επί τη βάση λοιπόν της δικής μου εισαγωγής όπου εντόπισα αυτά που σήμερα ε, είναι και τα θετικά σημεία αλλά και τα κρίσιμα σημεία της εφαρμογής αυτής της υλοποίηση αυτής θεωρήσαμε σωστό σήμερα να γίνει μια παρουσίαση των τριών αυτών μελετών που ζητήσαμε το πρώτο δημιουργική Ευρώπη, πολιτισμική Ευρώπη υπότιτλος αφιερώνεται σε θέματα πολιτισμού το διαχειρίστηκε η θεματική, το θεματικό τμήμα Β η κυρία Λάτζαρο από το Πανεπιστήμιο του Ουτρέχτης στην οποία ευχαριστούμε. Δεύτερη μελέτη. Αλλά μοντου που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, είναι σημείο αναφοράς για όλους και τον ευχαριστούμε που είναι σήμερα μαζί μας. Μια ενδελεχής ε, μελέτη για το ίδιο θέμα της Δημιουργικής Ευρώπης, σε ένα ενδιάμεσο χρονικό σημείο εφαρμογής επί τη βάση ενός ερωτηματολογίου που είχε υποβληθεί στο Creative Desk από τον κύριο Μοντό και την κυρία Αλμαντετέ και θα το προσθέσει ο κύριος Μοντό. Δηλαδή, η τρίτη μελέτη είναι μια αξιολόγηση της Δημιουργικής Ευρώπης που έγινε in-house από το Γραφείο Μελετών του Κοινοβουλίου το οποίο εκπροσωπεί ο θαυμάσιο αυτό ερευνητή που, που έχω δίπλα μου. Και ίσω ε, στο τέλος παρουσίασή σα ε, μπορεί να πω και εγώ δύο λόγια για να θυμίσω και τα σημεία πολύ σύντομα που είχαμε υπογραμμίσει σημειώσει την περασμένη φορά, στην προηγούμενη συνεδρίαση. Και από εκεί πέρα θα ε, υπάρξουν και ερωτήσεις σε συζήτηση με τα μέλη για περαιτέρω συζήτηση. Θα δώσω το λόγο πρώτο στους κοιόδης και μετά στους ενδιαφερομένους. Και μετά ελπίζω ότι ε, θα είναι η σειρά της Κομισιόν που θα ακούσουμε την άποψή της με ενδιαφέρον. Θα δώσω το λόγο στην πρώτη ερευνήτρια. Ζητώ να μείνετε όλοι στα 10 λεπτά ο καθένας. Έχουμε και διαφάνειες. Νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει. Παρακαλώ. Η κυρία Λάτζερο. αυτή ήταν η σειρά που είχε προταθεί. Να ξεκινήσουμε από τα PRS. Εντάξει. Όπω όπως θέλετε. Καμία αντίρρηση. Good afternoon. Καλησπέρα. Καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Κώστα που μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την εσωτερική ανάλυση μας ε, ως εισαγωγή. Είναι η Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση ε, για την Εφαρμογή που έφτιαξε το EPRS. Είναι ε, η καθημερινή δουλειά που κάνει το EPRS για τέτοιες εκθέσεις εφαρμογής από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ε, προσπαθούμε ταυτόχρονα να κάνουμε μία ανάλυση η οποία στην ουσία λαμβάνει υπόψη ότι το ε, Creative Europe, Δημιουργική Ευρώπη, υπάρχει εδώ και τρία χρόνια. Όταν έγινε η πρώτη μελέτη δεν μπορούσαμε να έχουμε μια πλήρη αξιολόγηση, όμως τώρα ε, μπορέσαμε να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να συλλέξουμε τις πληροφορίες οι οποίες ε, θα μας επιτρέψουν αργότερα μια καλύτερη ανάλυση. Εδώ βλέπετε και διάφορα άλλα είδη αναλύσεων που έχουμε κάνει, την ε, μονάδα αξιολόγησης επιπτώσεων EXPOST. Ε, από την μονάδα αυτή λοιπόν έχουν δημιουργηθεί αυτές οι εκθέσεις που βλέπετε στην οθόνη. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν κάποιες αξιολογήσεις του Creative Europe, υπάρχει και ο κανονισμός ε, επί του οποίου βασίζεται η Δημιουργική Ευρώπη. Το 2013 υποστηρίχθηκε ο κανονισμός από μία μελέτη επιπτώσεων η οποία υπογράμμιζε τις, τα πιθανά πλεονεκτήματα που θα είχε μια ολοκλήρωση ε, των προηγούμενων προγραμμάτων του Culture και του Media και μια συγχώνευσή τους. Επίσης, δόθηκε προσοχή στα πλεονεκτήματα που θα είχε ένα οικονομικό ε, μέσο, ένα χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο θα θα είχε εφαρμογή σε όλους τους ε, τομείς, ε, κάτι που παραδοσιακά ήταν δύσκολο στο παρελθόν, ε, γιατί δεν υπήρχε υποστήριξη από το κοινό. Επίσης υπήρξε μια διάμεση αξιολόγηση για τα δύο προγράμματα, το Culture και το Media, Ξεκινώντας λοιπόν με την ενδιάμεση αξιολόγηση του culture, πολιτισμός, πέρα από τα θετικά στοιχεία που υπογραμμίστηκαν, μεταξύ των οποίων και η συμβολή στην διασυνοριακή συνεργασία, υπήρξε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε καλύτερα με κριτικό πνεύμα ε, την έλλειψη ε, επιτευγμάτων ως προς την ψηφιοποίηση. Το ίδιο ε, ισχύει και για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Media. Εκεί υπήρξαν κριτικές περισσότερο προς την κατεύθυνση της ε, κατάλληλης αντίδρασης στην καινοτομία. Δεν υπήρχε κάποια εγγύηση ότι θα επιτευχθεί αυτό. Αφήστε με τώρα να αφιερώσω λίγα λεπτά στα συγκεκριμένα στοιχεία της ανάλυσής μας. Αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς που συνεισφέρει και στην ολοκλήρωση της εφαρμογής, της έκθεσης εφαρμογής, ε, για την οποία θα υπάρχει σήμερα ανταλλαγή απόψεων. Νομίζω ότι ε, επίσης ε, θα συμπληρωθεί και η δουλειά του συναδέλφου ε, Πόλα από τη γενική, αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά του προγράμματος, τα οποία θέτουν κάποιες προκλήσεις για το μέλλον. Κάποια, ε, λοιπόν, είναι πιο σημαντικά για τη συζήτησή μας σήμερα. Ξεκινώντας λοιπόν με μια υπενθύμηση να πω το ότι υπήρξε μια νέα δομή στο Creative Europe, ε, δηλαδή ε, το ότι υπήρχαν δύο κατευθύνσεις οι οποίες ε, μαζί συγχωνεύτηκαν και δόθηκε και μια τρίτη διάσταση, ένα χρηματοδοτικό μέσο που άπτεται όλων των θεμάτων, στην ουσία μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης και αυτή την αυξημένη κατάτμιση της αγοράς. Επίσης, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και την πρόκληση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και τις συνεχείς δυσκολίες που υφίστανται ως προς την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ειδικά για όσους βρίσκονται στη δημιουργική βιομηχανία, στον τομέα του πολιτισμού. Σε στατιστικό επίπεδο, ε, στον τομέα του πολιτισμού, <clears throat> υπήρξε συλλογή στοιχείων, δεδομένων, παρόλο που υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί. Και μπορέσαμε να εκδώσουμε μέσω της Eurostat νέες στατιστικές για τον πολιτισμό, και ε, μελέτες που βασίστηκαν στην έκθεση για τον πολιτισμό ΙΣΝΕΤ, το Ευρωβαρόμετρο και την έρευνα της Eurostat για τον ε, προϋπολογισμό των οικοκυριών. Όλα αυτά μας βοήθησαν να συλλέξουμε και στατιστικές σε επίπεδο περιγραφικό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Creative Europe που υποβλήθησε συζήτηση και θα συζητηθεί και στο μέλλον, είναι η δημιουργία του νέου χρηματοδοτικού μέσου, της νέας διευκόλυνσης ε, εγγύσεων, ε, το οποίο θα υπάρχει στο μέλλον με κάποια καθυστέρηση βέβαια. Μια καθυστέρηση η οποία δικαιολογείται βέβαια από τις ε, δυσκολίες του να προσελκύσει επενδυτές σε έναν τομέα όπου τα έσοδα και τα κέρδη δεν μπορεί κανείς ε, να τα απολαύσει άμεσα. Τα στοιχεία που θα σας δώσουμε σήμερα επίσης θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε σε πρώτη φάση την ενδιάμεση αξιολόγηση της Creative Europe που θα δώσει η Κομισιόν μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. Θα τελειώσω με τα πέντε σημεία που φαίνεται ότι είναι κρίσιμα, όχι απαραίτητα αρνητικά, αλλά ε, και για την ε, θετική, για την ε, καλή λειτουργία του Creative Europe. Πρώτον, έχουμε την ενσωμάτωση και ολοκλήρωση και συγχώνευση όλων των προγραμμάτων που είχαμε στο παρελθόν, τα οποία ήταν χωριστά. Στην ουσία υπάρχει και μία ε, ολοκλήρωση και συγχώνευση και των υπηρεσιών της Κομισιόν που δεν είναι απαραίτητα μόνο στο επίπεδο της διαχείρισης αλλά ενέχει και προκλήσεις ε, λόγω της διαφορετικής θέσης στην αγορά των δύο αυτών τομέων στους οποίους επενδύει το πρόγραμμα. Είναι δύο τομείς που απευθύνονται σε διαφορετικές αγορές και διαφορετικές αποτυχίες, αστοχίες της αγοράς. Ο ρόλος επίσης ε, των ε, σταθμών ε, της Δημιουργικής Ευρώπης, τα Creative Europe Desks, CEDs, ο ρόλος και η δράση τους σε πολλές περιπτώσεις ήταν περισσότερο πληροφορικός, πληροφοριακός. Όμως θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν καταλήτη ε, για να, μπορούν, να μπορέσουμε να χαρτογραφήσουμε τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ειδικότερα της βιομηχανίας, ε, του πολιτισμού και της δημιουργίας. Τώρα, η λογική της επέμβασης και η ανάγκη εγγύησης μιας ε, συγκεκριμένης οικονομικής γάμας σε έναν τομέα όπου υπάρχει περιχαράκωση ως προς το χρηματοδοτικό ε, θέμα. Ε, υπήρξε μια σειρά από υποστηριζόμενα σχέδια Και αυτό θα γινόταν μόνο εφόσον υπήρχε εγγύηση για την αποδετικότητα αυτών των σχεδίων ε, κατά την έναρξη του προγράμματος. Ένα θέμα το οποίο ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο για μένα προσωπικά, λοιπόν, διότι μπορεί να μας ε, οδηγήσει στη γενικότερη αξιολόγηση του προγράμματος γενικότερα, είναι το σύστημα των δικτών με το οποίο έπρεπε να συνοδεύεται το πρόγραμμα εξ αρχής, από τη δημιουργία του. Αυτοί οι δείκτες, από τον κανονισμό ήδη, φαίνεται ότι ήταν λίγο πιο προαιρετικοί και τελικά δεν έχουν γίνει πλήρως ε, λειτουργικοί, οπότε ε, δεν έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που θα αντικατοπτρίζει καλύτερα τους στόχους του προγράμματος για να έχουμε ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα που θα παρακολουθεί όλες τις ε, δραστηριότητες και δομές μέσω των οποίων λαμβάνει η χώρα το πρόγραμμα. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο το οποίο δεν αφορά μόνο και απαραίτητα την Δημιουργική Ευρώπη, το Creative Europe, είναι λίγο πιο γενικό, έχει να κάνει με την υποστήριξη του κοινού γενικότερα. Και σε αυτή την περίπτωση πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τη δυνατότητα εγγύησης ταυτόχρονα και την ίδια στιγμή μιας ποικιλομορφία στον τομέα της δημιουργίας και του πολιτισμού ε, σε συνδυασμό με μια ανταγωνιστικότητα. Πρέπει και τα δύο στοιχεία αυτά να υποστηρίζονται λοιπόν. Ε, θα σταματήσω εδώ και μετά με τη χαρά μου θα συνεχίσω αν χρειαστεί. Ευχαριστούμε πολύ για τον πολύ συνοπτικό τρόπο με τον οποίο κάνατε την παρουσίαση και την ανάλυση σας. Να σας ε, διαβεβαιώσω ότι επειδή έχει λίγη ε, ζέστη θα ανάψουμε το air condition οπότε σύντομα θα αισθανόμαστε όλοι καλύτερα. Τώρα δίνω το λόγο στον ε, καθηγητή Λάτσαρο. Στην καθηγητρία Λα... κυρία Λάτσαρο. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης που με προσκάλεσε να παρουσιάσω τη μελέτη που συμπίλησα για την Επιτροπή για τη Γενική Διευθυντική πολιτική. Πρόκειται λοιπόν για τη μελέτη σχετική με την υλοποίηση της νέας Δημιουργικής Ευρώπης, το υποπρόγραμμα για τον πολιτισμό συγκεκριμένα. Και θα σας ενημερώσει και ο συνάδελφος για το τμήμα που αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε λίγο χρόνο. Σας καλώ λοιπόν να μελετήσετε, να κοιτάξουμε πολύ γρήγορα την μελέτη η οποία έχει δι... διτεθεί στο διαδίκτυο και να περάσουμε στα συμπεράσματα λίγο πολύ. Ιδιαίτερα θέλω να τοποθετηθώ στο υπόβαθρο του στόχους το πεδίο που κάλυψε αυτή η μελέτη. Θα παρουσιάσω τα κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα και βέβαια συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως. Ανεφέρθη ήδη το υπόβαθρο. Δηλαδή ένα νέο πλαίσιο του προγράμματος Creative Europe που όπως ξέρετε συγχωνεύει τον πολιτισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα δύο αυτά υποπρογράμματα ε, που γίνονται το νέο Creative Europe με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας. Το culture και το media ξέρετε ότι υπάγονται σε δύο διαφορετικές γενικές διευθύνσεις, την ΕΑΚ e και την Connect, αντίστοιχα για τον πολιτισμό και τα μέσα. Έτσι λοιπόν η μελέτη μας στόχο έχει να σας εξηγήσει πώς προχώρησε η υλοποίηση των υποπρογραμμάτων, Ποια ήταν τα κύρια μελήματα που αντιμετώπισαν οι ετούντες και οι πληθέντες να υλοποιήσουν τα προγράμματα, εκείνοι δηλαδή που είναι οι κύριοι χρήστες. Στόχος μας ήταν μια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στηριζόμενη σε μια έρευνα από, τα, ε, από τις υπηρεσίες του Creative Europe με πρώτες εντυπώσεις και ένα διαδικτυακό, διαγραμμικό ερωτηματολόγιο με ένα πρόγραμμα σχετικό με την εξέταση της υλοποίησης. Ξέρετε, αυτά τα Creative Europe Desks αποτελούν το σημείο συνάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του τελικού χρήστη και του κράτους μέλους. Γι' αυτό επελέγησαν, γιατί έχουν μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα και μπορούν να αξιολογήσουν ε, πώς προχωράει η κατάσταση. Έχουν μια πολύ σημαντική προοπτική λοιπόν και ταυτόχρονα επειδή δεν είχαμε και απεριόριστο χρόνο στη θέση μας, θεωρήσαμε ότι η επιλογή αυτών των ε, γραφείων εξυπηρέτησης ήταν η καλύτερη για να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν ότι οργανώσαμε ένα διαγραμμικό ερωτηματολόγιο. Θα το δείτε στο παράρτημα της μελέτης, οργανωμένο σε έξι τμήματα, όπου ζητούμε το προφίλ του γραφείου ενημέρωσης, τις προτεραιότητες, γενικούς στόχους, ε, δικαιούχους και πληροφορίες σχετικές με αυτούς, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αλλαγές σε σχέση με το Culture 2007-2015 και άλλες γενικές παρατηρήσεις. Είχαμε και ε, κλειστές ερωτήσεις, δηλαδή πολλαπλές επιλογές και ανοιχτές στο ερωτηματολόγιο. Πολύ σύντομα τα αποτελέσματα, τα κύρια ευρήματά μας ήταν ότι καταρχάς είχαμε ευρή ανταπόκριση, σημαντική στατιστικά, από 32 γραφεία εκ των 39 υφισταμένων γραφείων ενημέρωσης, άρα έχουμε καλή κάλυψη σε παιδοκρατών μελών και λοιπόν κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης, το υποπρόγραμμα για τον πολιτισμό του Creative Europe θεωρείται πολύ σημαντικό, κρίνεται ως πολύ σημαντικό για τον πολιτισμό στην Ευρώπη και τις λοιπές χώρες, έχει μεγάλη σημασία. Τα περισσότερα από τα γραφεία ενημέρωσης μας λένε ότι είναι επιτυχής η υλοποίησή του και σε σχέση με τους στόχους του ίδιου του υποπρογράμματος, αλλά και σε σχέση με τους γενικούς στόχους ε, του Creative Europe. Και οι ε, φορείς πολιτιστικοί κρίνουν θετικά από ό,τι ε, μας λένε στα ερωτηματολόγια. Κάποιες ε, προτεραιότητες μόνο εξετάζουν με πιο επικριτικό βλέμμα από ότι κάποιες άλλες, θα δούμε μετά ποιες. Το κόστος είναι ο κύριος φραγμός σε σχέση με την υλοποίηση, δηλαδή δημοσιονομικά ζητήματα. Οι μικρές, μικρο και μεγαλύτερες οργανώσεις και τομείς όπως η αρχιτεκτονική, το σχέδιο, οι φυρμοσμένες τέχνες, τα οπτικά, ακουστικά και η πολιτιστική κληρονομιά έχουν τη μικρότερη εκπροσώπηση σε δικαιούχους. Η εμπειρία είναι κύριο κίνητρο, ενώ ταυτόχρονα τα οικονομικά είναι το κύριο εμπόδιο για συμμετοχή σε προγράμματα. Ε, που βλέπουμε την καλύτερη εφαρμογή, που βλέπουν ε, τα εθνικά γραφεία ενημέρωσης ε, την καλύτερη εφαρμογή. Ε, στην προαγωγή λοιπόν της ε, διεθνικής κινητικότητας καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού, προαγωγή πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, οικοδόμηση δυνατοτήτων, ανάπτυξη ευρωπαϊκής πλατφόρμας, ευρωπαϊκών πλατφορμών, ε, παραγωγή καλλιτεχνικού ή πολιτιστικού προϊόντος, έργου, παραγωγή ε, ισχυρών και διαρκών εταιρικών σχέσεων μεταξύ συντονιστών και συνδιοργανωτών. Δηλαδή μια ευρωπαϊκή συνεργασία θεωρείται το καλύτερο συστατικό για την επιτυχία ενός χρηματοδοτούμενου έργου. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής και στράτευσης ε, των οργανώσεων που εμπλέκονται. Αυτά είναι τα θετικά λοιπόν μέχρι τώρα στην εφαρμογή του προγράμματος. Τα αρνητικά ή τα αδύναμα σημεία ήταν η αξιολόγηση, ο έλεγχος ολογιστικός δηλαδή, η αξιολογηση ο ελεγχος λογιστικος δηλαδη η υλοποιηση σε, διεθνές, σε διεθνικό επίπεδο των ε, επαγγελματικών δυνατοτήτων, ε, ο κίνδυνος ε, κανιβαλισμού, επανάληψης κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή διάκριση με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα και αυτό πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς και η υπηρεσία να εξετάσουν, αλλά βέβαια και τα εθνικά γραφεία. Η υποστήριξη κυκλοφορίας προαγωγής, μετάφραση ευρωπαϊκής ε, λογοτεχνίας, το θέμα δηλαδή της, ε, γλωσσικής, της ε, λογοτεχνικής μετάφρασης, προαγωγή της γλωσσικής πολυμορφίας, δυστυχώς, η διάδοση έργων των αποτελεσμάτων αυτών και των επιτευγμάτων τους και ισορροπία μεταξύ καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων. Ε, συστάσεις λοιπόν πολύ σύντομα για να καταλήξουμε. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει προτεραιότητες και άλλες πτυχές που έχουν τη μεγαλύτερη επιτυχία στην υλοποίηση, όπως ανέφερα νωρίτερα, να διευκολύνει να επανεξετάσει προτεραιότητες και άλλες πτυχές που φαίνεται να έχουν λιγότερο η επιτυχία στην υλοποίησή τους, να περιορίσει το δυσανάλογα περιορισμένο αριθμό ε, μάλλον τη δυσαναλογία στα νούμερα των δικαιούχων και των ετούντων, άρα θα πρέπει και να ενισχυθεί ο προπολογισμό ε, για να υπάρχει και καλύτερη, μεγαλύτερη συμμετοχή δικαιούχων και καλύτερη εκπροσώπηση όλων των τομέων πολιτιστικών και δημιουργικών. Ε, περισσότερη υποστήριξη να δοθεί σε έργα μικρού, μικρής κλίμακος, να κοινοποιούνται περισσότερο και ευρύτερα οι ιστορίες ε, εκείνων που επέτυχαν και να διευκολύνει βέβαια η ανταλλαγή της τεχνογνωσίας, ε, η ε, παγίωση των βελτιώσεων που εξασφαλίζονται σε κάποια προγράμματα, κυρίως όσον αφορά την υλοποίηση και την απλούστευση της λειτουργίας των προγραμμάτων και βέβαια για να ολοκληρώσω να ενσωματωθούν περισσότερο αυτά τα εθνικά γραφεία στη διαδικασία των εισλήψεων αποφάσεων και κυρίως μια καλύτερη συμμετοχή και επικοινωνία των, στα δεδομένα και τις πληροφορίες ε, σε θέματα πολιτισμού και μέσων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την καθηγήτρια. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν να φτάσετε σε μία σύνοψη σε λίγα λεπτά, για λίγα λεπτά μάλλον, δεδομένης λεπτομέρειας τέθησαν, υπευλήθησαν και πάρα πολλές ερωτήσεις ε, και θα υπάρξουν φαντάζομαι ε, στην επόμενη φάση. Ο κύριος Μοντό τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω λίγα γαλλικά. Ε, θα υποφεληθώ από τις διευκολύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια, η παρουσίασή μου είναι στα αγγλικά, στο PowerPoint. Δεν θα αναφέρω όλα τα ζητήματα που ήδη ανέφεραν οι συνάδελφοι σχετικά με το χρόνο που χρειάστηκε για να γίνει αυτή η μελέτη. Θα μιλήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται σχετικά με το πλαίσιο, τη μεθοδολογία, τα πρώτα ε, αποτελέσματα ε, των ε, διαγωνισμών και τα διάφορα αποτελέσματα των ερευνών καθώς και τα συμπεράσματα. Λοιπόν, το πρώτο που καταφέραμε να κάνουμε ήταν να κατανοήσουμε ποια ήταν η σχέση αυτού του προγράμματος με το προηγούμενο που πήγε μέχρι το 2014 όπου ξεκίνησε το καινούριο που ήταν το Culture Media και Media Mundus. Ε, το ε, ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να δημιουργήσει μια κουλτούρα για να υποστηρίξει τα οπτοκουστικά μέσα, τα ντοκιμαντέρ, τα video games, τα φεστιβάλ, τα δίκτυα των κινηματογράφων. Όλα αυτά αποτέλεσαν μια καινοτομία για το διαπολιτισμικό πρόγραμμα που θέλαμε να προωθήσουμε. Ζητώ συγγνώμη, έχω ένα πρόβλημα με την παρουσίαση, λέει ο μιλητή. Voilà, euh, euh, Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές ε, που έχουν γίνει. Είχαν να κάνουν ε, ε, βασικά υπήρξε μια επανάληψη των βασικών ε, στοιχείων. Βέβαια υπήρχαν και κάποια στοιχεία που εγκαταλείψαμε όπως τα πιλωτικά προγράμματα και το I2I που έχει να κάνουν με την παραγωγή. Αλλά προσθέθηκαν νέες γραμμές όπως η ανάπτυξη του κοινού, τα κονδύλια για την συμπαραγωγή και τα κονδύλια για το Ταμείο Εγγύησεων. Αυτές ε, οι αλλαγές οδήγησαν σε νέους ε, εποφελούμενους ε, και όσον αφορά στην ανάπτυξη του κοινού και την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης του περιεχομένου. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι η ίδια που ακολούθησε και η Ελιζαμπέτα. Εμείς στην ουσία επικεντρωθήκαμε στα Media Desk Στείλαμε ένα εντελώ ανώνυμο ερωτηματολόγιο, δηλαδή στο τέλος της έρευνας ε, δεν ξέραμε παρά μόνο με κάποιους ε, που είχαν αναφέρει συγκεκριμένε καταστάσεις στη χώρα τους, δεν ξέραμε ποιος είχε απαντήσει. Αυτό το χρειαζόμασταν για να ε, κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ του εκτελεστικού οργάνου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε 32 απαντήσεις, όμως υπάρχουν κάποια media desk που καλύπτουν πολλές χώρες όπως τη Γαλλία, την Ισπανία, ή πολλές ε, περιοχές μάλλον στις αντίστοιχες χώρες, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και είχαμε είτε τη χώρα που απαντούσε είτε τα media desk αυτής της χώρας. Είχαμε 32 λοιπόν απαντήσεις οι οποίες κάλυπταν 83,35% των media desk. Υπήρχαν και κάποια που δεν μπόρεσαν ποτέ να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, το οποίο γενικά φορούσε τρεις ομάδες ερωτήσεων της ε, σχέσεις ε, μεταξύ της Επιτροπής και των γραφείων, πώς ε, διαχειριζόμαστε την αλλαγή και ποια είναι τα βασικά εργαλεία που χρειάστηκαν οι ε, ε, συμμετέχοντες, τα πρώτα αποτελέσματα και τις προτάσεις που έκαναν τα Media Desk. Είχαμε 240 σελίδες ε, απαντήσεων που είναι στο παράρτημα της έκθεσής μας για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Τα πρώτα αποτελέσματα τώρα, μετά από δύο χρόνια, με τους διάφορους διαγωνισμούς που έγιναν, συλλέχθησαν βάσει των δεδομένων που είχαμε από το site του Creative Europe. Αυτή τη στιγμή έχουμε μερικά αποτελέσματα, αλλά από αυτά παίρνουμε ε, πολλές πληροφορίες. Πάνω από 800 φάκελοι έχουν κατατεθεί ε, και παρόλο που όλες οι προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν ήταν ε, online, ε, έχουμε όλα τα στοιχεία. 1.800 λοιπόν φάκελοι κατατέθηκαν στη γραμμή διανομή, ε, στο θέμα ε, διανομής, ανάπτυξης κτλ. Και τα αποτελέσματα που βλέπετε εδώ στον πίνακα στην ουσία μας δείχνουν τη σύγκριση μεταξύ των υποψηφιωτήτων αναχώρα, όποιος και αν ήταν ο τομέας, και ε, του αριθμού των σχεδίων που υποστηρίχθηκαν, που επιλέχθηκαν μετά από τη διαδικασία επιλογής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πέντε χώρες ε, που είναι πάνω από το 60% ε, για τα για τις υποψηφιότητες που είχαν. Μετά έχουμε μια σειρά χωρών που είναι γύρω στο 50% και μετά η βασική ομάδα χωρών που είναι κάτω από το 50% με κάποιες εκπλήξεις. Βλέπουμε ε, ότι οι δύο τελευταίες χώρες, ε, δυστυχώς κυρία Πρόεδρε, είναι η Ιταλία 26,2 και αμέσως από πάνω η Αγγλία 28,6. Η Γαλλία και η Γερμανία είναι και αυτές ε, σε αυτή την ομάδα των χωρών που δεν μπόρεσαν να επιλεγούν στον ίδιο βαθμό από το πρόγραμμα. Τα βασικά συμπεράσματα λοιπόν που μπορέσαμε να βγάλουμε και να κρατήσουμε ήταν οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. Ε, ποια είναι τα εργαλεία επίσης της Δημιουργικής Ευρώπης ε, και τέλος αυτό που έλεγαν τα Media Desk, οι διάφορες γραμμές υποστήριξης, οι τομείς. Τώρα, Όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ του οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή των Γενικών Διευθύνσεων, καταρχάς ε, αυτή η συγχώνευση ήταν μια πραγματική μάχη μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων, του οπτικο-ακουστικού ε, και του πολιτισμού. Εδώ βλέπετε ότι ε, αυτά τα παρουσιάζουμε ως συστάσεις, διότι έρχονται κατευθείαν από τα Media Desk. Υπάρχουν πολλά στοιχεία και έγγραφα που έχουν ε, θέσει στη διάθεσή μας τα Media Desk, όμως αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ από την Κομισιόν ή από τον οργανισμό για να υποφεληθούν όλοι. Πολύ συχνά στο ερωτηματολόγιο διάβαζα ότι κάποια νέα Media Desk είχαν χαθεί ως προς την εφαρμογή του προγράμματος. Talk to them, μιλήστε τους. Αυτό ήταν ε, η άποψη των Media Desk που στην ουσία, όπως σας είπα, δεν είχαν μπει στη λογική του προγράμματος ε, και δεν ε, αισθάνονταν ασφάλεια, οπότε ζητούν ενίσχυση της αλληλοπληροφόρησης μεταξύ των δύο μερών. Περισσότερες πληροφορίες επίσης για τις εφαρμογές και που επέτυχαν και που απέτυχαν. Αυτό ε, είναι μια μεγάλη διαφορά, ε, διότι τα Media Desk είχαν ε, στην ουσία τη δυνατότητα να εξηγήσουν ποιες ήταν οι επιλογές τους και γιατί τις έκαναν. Επίσης, χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στις αξιολόγηση και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, όπως και στη διαδικασία επιλογής, καλύτερη συνεργασία μεταξύ ε, αυτών των media desk για να μπορέσει να υπάρχει ανταλλαγή πρακτικών, των πρακτικών και πληροφορίων. Επίση, δεν υπάρχει οργανόγραμμα του οργανισμού και δεν μπορεί που να είναι δημόσιο και δεν μπορεί κανεί να επικοινωνήσει σωστά, δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, σε ποιο email. Και ε, θέλουν και περισσότερε συναντήσει και online με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον πήγα λίγο γρήγορα, λέει ο μιλητή, αλλά θα πάω ακόμα πιο γρήγορα. Les outils, les outils globalement. Τα γενικά εργαλεία είναι αρκετά ικανοποιητικά, όμως ε, το πόρταλ είναι πολύ περίπλοκο και πρέπει ε, να βελτιωθεί. Επίσης, ε, η online επικοινωνία είναι ικανοποιητική. Οι εφαρμογές παραμένουν περίπλοκες. Υπάρχουν πέντε διαφορετικοί οδηγοί. Υπάρχει πολύ μεγάλη ορολογία και οι διαφορετικές προσεγγίσεις της Κομισιόν, του Οργανισμού και των οδηγών. Επίσης υπάρχει και το σύστημα της αυτόματης απάντησης που και αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Ε, τώρα, οι γραμμές υποστήριξης, οι τομείς, ε, ε, δεν θεωρείται ιδιαίτερα ευέλικτο το πρόγραμμα και χρειάζεται περισσότερη ποιότητα στο point system. Ε, ένα θέμα που έθεσαν πολλά media και και τα πολύ μεγάλα και τα πολύ μικρά. Αυτό το σύστημα των αυτόματων ε, πόντων ε, κάπως δίνει ένα προνόμιο στις μικρές χώρες στο επίπεδο programming Έχουμε κάποιους πόντους για τις μικρές χώρες ε, και πέντε πόντους για το σύστημα ε, νέων. Οπότε από αυτό το σύστημα, από ό,τι φαίνεται, θεωρητικά εποφελούνται οι μικρές χώρες, όμως τα αποτελέσματα που είδαμε στον πίνακα δείχνουν ότι οι μεσαίες χώρες τελικά έχουν περισσότερο η καλύτερη θέση. Ε, γενικά υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος ε, ε, είναι κάπως στρεβλός και έχει στρεβλά αποτελέσματα και αποτελέσματα που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Το βασικό θέμα λοιπόν που τέθηκε για τις γραμμές υποστήριξης ήταν η δυνατότητα για crossover projects που είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Το πρώτο συμπέρασμα, πολύ γρήγορα, το πρόγραμμα θεωρείται ότι έχει ανταποκριθεί στις γενικότερες ανάγκες του τομέα και σε νέες ανάγκες. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια ιδιαίτερα περίπλοκη και μεγάλη διάρθρωση, επεκτεταμένη διάρθρωση, παρόλο που υπάρχουν βελτιώσεις. Το θέμα της διάρκειας επίσης των αξιολογήσεων που έγιναν μέσα στα πλαίσια του προγράμματος φαίνεται ότι ότι ε, ε, είναι πολύ μεγάλες ε, οι περίοδοι, ενώ ας πούμε στο Eurimages έχουμε 7 εβδομάδες μόνο. Τώρα, για το γενικότερο προϋπολογισμό του προγράμματος Creative Europe υπάρχουν όλο και περισσότερες χώρες, όλο και περισσότερα αιτήματα και επαγγελματίες, άρα ε, βλέπουμε ότι αυτό δεν συνάδει με, με τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός δεν αυξάνεται ανάλογα με τις ανάγκες και ε, δεν είναι ευχαριστημένοι συμμετέχοντες γιατί υπάρχουν πολλές απορρίψεις. Αυτό ήθελα να πω πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Σας ευχαριστώ. Είχαμε λοιπόν τρεις, τρεις φωτογραφίες, απεικονίσεις πολύ ενδιαφέρουσες και ως προς τις θεματικές τους αλλά πέρα από τις παρουσιάσεις PowerPoint έχετε στη διάθεσή σας των μελετών, των κειμένων και μπορείτε ενδελεχέστερα να εξετάσετε όλα αυτά. Να ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους τους ε, συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Κοιτάω και το χρόνο για να δω πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε 15 λεπτά κατά μέγιστον. Θα επιφυλαχθώ εγώ να πω ένα-δύο λόγια στο τέλος. Σημειώνει η γραμματεία. Απλώς ε, ε, να σας πω δύο ημερομηνίες σκέτες, λέει η πρόεδρος. Είχαμε πει στους επιτρόπους, είχαμε επαναλάβει ότι παρά την έμφαση και στην πρόσφατη σύνοδο και γενικώ ε, εκφράζεται από διάφορους επικεφαλής κυβερνήσεων και ελπίζω και από την Κομισιόν, έχουμε θέσει σε πιο κεντρικό ε, πλαίσιο ε, για την ενδιάμεση αναθεώρηση ε, μια η σημαντική ενίσχυση των πόρων αυτών των θεματικών και να σας δώσω το εξής δεδομένο. Ο δείκτης επιτυχία των πράγμα των, των πολιτιστικών ε, λέγει 20% αλλά σε κάποιες γραμμές και σκέφτομαι τη συνεργασία γιατί εκεί θα συγκλίνουν όλα αυτά έχουμε δείκτη 11% ε, και μιλούμε για ένα τομέα ο οποίος ε, απεδείχθη ανθεκτικός και πάρα πολύ ενεργητικός και μιλούμε για τα μίντια που έχουν το 56% συνολικά του προϋπολισμού ως θεματική και έχουν και μια αυξημένη ικανότητα αν θέλετε ανταπόκρισης αλλά και εκεί είμαστε σε ένα 43% ε, μέσου όρου ε, ανταπόκρισης στα προγράμματα. Αυτά είναι ξερά μεγέθη. Το είχα πει και στην εισαγωγή, αυτό υπάρχει αυτή η βαθμολογία, το σύστημα της βαθμολογίας, το point system. Υπήρξε και μια πρόταση κανονισμού και από πλευράς Κοινοβουλίου για να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών. Αυτή η αυτόματη μέθοδος όμως ε, κινδυνεύει να στρεβλώσει, αν θέλετε, την πραγματικότητα της πολιτικής παραγωγής στην Ευρώπη. Και αυτό το λέω και προς την Κομισιόν, πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το θέμα της βαθμολογίας που πολύ συχνά είναι υπερβολικά άκαμπτη. Να μην προσθέσω άλλα, γιατί το έκανε στην εισαγωγή μου. Να δώσουμε το χρόνο συνεδρίφωση που δεν είχα μιλήσει και την προηγούμενη φορά. 1,5 λεπτό καθένα παρακαλώ. Ξεκινάω από αυτούς που ζήτησαν ήδη το λόγο, ε, η κυρία Εβερτ, Κάμερ Εβερτ, Βέιντα, Σοϊντρόβα, Βουέρτ Μόργανο και Εύανς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και έτσι θα είμαι σύντομη. Νομίζω ότι θα πρέπει ιδιαίτερα να μας απασχολήσει ο τρόπος της αξιολόγησης. Βεβαίως τα δύο προγράμματα πολιτισμός και μέσα έχουν ε, συνενωθεί. Πρέπει πάντως να μεριμνούμε έτσι ώστε οι συνεργατικές αυτές ε, δράσεις, η συνεργατική τους παρουσίαση να είναι πιο ορατή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι. Δεύτερον, δεν μπορούμε να επιλέγουμε και να υποστηρίζουμε μόνο τα μεγάλα ε, προγράμματα αντί για τα μικρότερα. Ε, μεγάλο πρόγραμμα άλλωστε δεν σημαίνει και περισσότερη ορατότητα στο κοινό. Ε, πιστεύω ότι υπάρχει άλλωστε και πρόβλημα διαφάνεια ω προς την επιλογή των προγραμμάτων. Πολλέ φορές δεν είναι κατανοητό πώς κατανέμονται οι πόντοι, με ποια βάση, τι είναι αυτό το οποίο οδήγησε σε μια θετική ή σε μια απορριπτική απόφαση. Και εδώ χρειάζεται λοιπόν περισσότερη δουλειά. και βεβαίως στο πρόγραμμα για τον πολιτισμό πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο δημιουργικό έργο. Αν και ο παραγωγικός ε, τομέας του πολιτισμού φαίνεται κάπως να υποχωρεί. Γι' αυτό λοιπόν ίσως θα μπορούσατε με βάση και τις δικές μας τις εμπειρίες, τις δικές σας εμπειρίες να μας πείτε εάν η κλασική εκδοχή, ο κλασικό τομέα του πολιτισμού και ο καλλιτέχνης κινδυνεύουν να μείνουν πίσω γιατί ιδιαίτερα προάγεται το δίκτυο και η δικτύωση των ε, καλλιτεχνών. Βεβαίω είναι πολύ καλά και σημαντικά τα ε, δίκτυα, αλλά πρέπει να εξασφαλίσετε μια ε, αηφορία στη δουλειά αυτή. Ευχαριστώ πολύ, Βέντα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω λίγο πολύ τα ίδια με τη συνάδελφο. Ευχαριστώντας βέβαια ε, εξ αρχής τους συναδέλφους ε, προσκεκλημένους για τη δουλειά τους. Εγώ είμαι σκιώδης ηγητής και ως εκ τούτου θα ήθελα να τοποθετηθώ για τη συγχώνευση των δύο αυτών πτυχών του πολιτισμού και των μέσων ε, μαζί των πολυμέσων γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη ε, ένας καλύτερος συνδυασμό των τομέων αυτών, μια καλύτερη συνεργασία. Η υποστήριξη για το πρόγραμμα Media επίσης. Και ε, τα προβλήματα στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων που επισημάνατε. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικά και πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις μικρότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε η υποστήριξη που τους προσφέρεται ε, να αντικατροπτίζει και την πολιτιστική πολυμορφία. Κυρία Ζόητροβα, ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω και εγώ στα όσα είπαν οι συνάδελφοι για το πρώτο ερώτημα και κυρίως τι σημαίνει και τι προσθεμένη αξία φέρνει η συγχώνευση των δύο αυτών τομέων μέσα στο πρόγραμμα Creative Europe. Δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη κατάσταση, δεν είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα και πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Δεν αποβαίνει βέβαια ε, προς όφελος της ε, χρηστής διαχείρισης των πόρων. Εάν αυτή η συγχώνευση περιπλέκει τα πράγματα και οργανωτικά και οικονομικά, που είναι πιο δύσκολο δηλαδή η διάθεση των κονδυλίων, τότε καλύτερα να τα χωρίσουμε και να είναι πιο απλά τα πράγματα, πιο κατανοητά για τον χρήστη, για την ε, μεθοδολογία επίση. Εσεί ε, μιλήσατε για την επικοινωνία σα με τα εθνικά γραφεία. Έχω πολύ καλή εμπειρία ε, στη συνεργασία με τα εθνικά γραφεία στην Τσεχική Δημοκρατία. Δεν με ξαφνιάζει λοιπόν το ότι είναι σε καλό επίπεδο οι δημόσιες δαπάνες. Ε, υπάρχουν ε, προγράμματα τα οποία μπορεί να είναι μικρότερα, πιο εύκολα διαχειρίσιμα, πιο προσβάσιμα για τον ενδιαφερόμενο. Σε αυτό θα συμφωνήσω και θα θέλαμε πιο πολλές πληροφορίες για να μπορούμε να αντιδρούμε πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Και έχω ακόμα και μια ερώτηση. Υπήρξε μια σύσταση για συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εσείς τι έχετε να προτείνετε. Εγώ πιστεύω ασφαλώς ότι χρειάζεται το λεγόμενο feedback, η διοχέτευση των στοιχείων και των πληροφοριών. Αλλά εσείς τι θα προτείνατε. Και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιαζόμαστε στις ε, μικρότερες προτάσεις, τα μικρότερα έργα. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τις ανταλλαγές πολιτιστικού περιεχομένου, ανταλλαγές μεταξύ ε, εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού και μην ξεχνάμε ακόμα και φύλακες ε, ε, ιστορικών μνημείων, παλατιών, κάστρων και το καθεξής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα. Το Σαββατοκύριακο συναντήθηκα με 150 καλλιτέχνες και αρμοδίους διαχείρισης πολιτιστικών προϊόντων σε ένα σχέδιο για τη συνεργασία για τον πολιτισμό από το οποίο είχα ξεκινήσει πριν από πέντε χρόνια και είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με αυτούς τους ε, ανθρώπους που κάνουν καταπληκτική δουλειά στη δημιουργία, στον πολιτισμό ε, για ε, λύσεις, ιδέες, προτάσεις και πάνω απ' όλα τη χρηματοδότηση. Και πρέπει να σας πω ότι το Creative Europe είναι η τελευταία τους λύση, η έσχατη λύση στην οποία θα καταφύγουν για χρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι και να τους υποστηρίξουμε και να τους ενημερώσουμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι ενσωματώνουν αυτό που συνιστά την Ευρώπη. Πρέπει το ε, όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι παρόν πάντοτε με λυπεί ιδιαίτερο το γεγονό ότι μόνο ως έσχατη θα στραφούν προ το Creating Europe. Ε, πρέπει αυτό να το λύσουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά ε, δημιουργικά έργα της Ευρώπης. Γιατί θα ε, πραγματοποιηθούν αυτά, θα υλοποιηθούν, μόνο που εμείς δεν θα είμαστε μέσα σε αυτά και αυτό θα ήταν κρίμα. Ευχαριστώ, Μόργαν. Κύριος Μόργαν, ε, ευχαριστώ. Ήθελα να ερωτήσω τον κύριο Ντόση ε, σχετικά με τους δείκτες που θεωρώ σημαντικό θέμα για το νέο πρόγραμμα. Ε, αυτοί οι δείκτες δεν είναι έτοιμοι, δεν είναι λειτουργικοί. Και επομένως υπάρχει ένα θέμα παρακολούθησης του όλου συστήματος. Και επομένω, πέραν τη ε, ανάγνωση παρουσίαση που κάνατε, πώ μπορείτε να μα πείτε κάτι σχετικά με αυτό και για την κυρία Λάτσαρο, ε, σχετικά με την ε, περιοδική, αν θέλετε, εξέταση των δικαιούχων. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε και ποια διαδικασία, αν θέλετε, ε, επανεξέτασης ή διόρθωσης υπάρχει, γιατί η δάλος με αυτή την περιπλοκότητα της βαθμολογίας ε, δεν πάμε πουθενά. Ε, επίσης, ανησυχώ ιδιαίτερα για την παρουσία του κυρίου Μοντού, όπου ταυτίζεται με τη θέση από ό,τι φαίνεται των Media Desk εκεί που μιλούμε για στρεβλωτικούς μηχανισμούς το οποίο είναι ιδιαίτερο ανησυχητικό. Αναφέρομαι σε θέματα διαφάνειας, σε θέματα πληροφόρηση επί των αποκλήσεων ε, και τη του κάποιων από τα στοιχεία αυτά. Μου φαίνεται ότι πέραν της οποιασδήποτε συγχώνευσης εδώ έχουμε ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα. Ε, ε, πάνω μας κρέμεται και το θέμα του προπολογισμού, για το οποίο δεν μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας αλλά είναι και αυτό στα υπόψη. Μάλιστα η κυρία Εύαν, λέει η πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω την κυρία Λάτζαρο επίσης για τα προγράμματα πολιτισμού με έκπληξη είδα ότι η πρόθεση της γλωσσικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας ήταν από τα πιο προωθημένα στην εφαρμογή. Τώρα εμείς γνωρίζουμε στην Επιτροπή πόσο ζωτική σημασία είναι όλα αυτά και πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τέτοια προγράμματα. Και ίσως αυτό να καλύπτεται στην έκθεση Fuller, αλλά μήπως μπορείτε να μας δώσετε μια ένδειξη σχετικά με την αιτία. Μήπως δηλαδή καλύπτει κάποιες ε, μειονοτικές ή περιφερειακέ γλώσσες στο πράγμα. Ευχαριστώ όλους. Στο σημείο αυτό θα στρεφόμουν στην ε, Κομισιόν ε, όπως και στον οργανισμό που είναι εδώ παρόντες. E και όπως ε, υπογράμμισαν και οι σκιώδεις, ε, είχαμε και εμείς πάρα πολλές ε, συναντήσεις με τους ενδιαφερομένους και με τα desk και με πάρα πολλούς οργανισμούς, ενώσεις, ενδιαφερόμενους φορείς ε, σε διάφορες χώρες, αλλά ιδιαίτερα στις χώρες των υποπρογραμμάτων. Παρακαλώ τους εκπροσώπους της ΕΑΣΙΕΑ και της Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε εκ μέρους τη ΔΕΛΤΑ Education and Culture. Έχουμε και τους συναδέλφους της Connect και του οργανισμού μετά, που θα μιλήσουν μετά από μένα. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, άρα δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες ε, για όλες τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία αυτή. Είναι πολύτιμες αυτές οι μελέτες και είναι και απολύτως έγκαιρες διότι τροφοδοτούν την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση σχετικά με το πρόγραμμα αυτό. Θα είναι λοιπόν πολύτιμο input ε, στη δουλειά που κάνουμε στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να βελτιωθεί το πρόγραμμα αυτό στο δεύτερο τμήμα, στην δεύτερη φάση, αν θέλετε, της λειτουργίας του. Ένα-δύο σημεία που ετέθησαν. Η ένταξη, η ενσωμάτωση του προγράμματος και τα θέματα που είχαμε τα τελευταία χρόνια παρά τις ε, εντάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από το γεγονός ότι έχουμε δύο διαφορετικές γενικές διευθύνσεις ε, επικεφαλής, είναι αμοιβαίως ε, εποφελές για όλους γιατί έχουμε μια ενιαία άποψη επί του ψηφιακού θεματολογίου και της ενιαίας αγοράς με μια πιο ε, πολιτιστική προσέγγιση αν θέλετε στην προάσπιση όχι μόνο των τεχνικών θεμάτων αλλά και των υπολείπων. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή συνολική εικόνα υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι εξακολουθούμε να διαχειριζόμαστε από κοινού το πρόγραμμα σε μια σταθερή βάση. Ο ρόλος των desk στο ε, σημείο στο οποίο έγινε αρκετή μνήμα και που συνεισφέρουν ουσιαστικότατα στις μελέτες. Είμαστε πολύ τυχεροί θα έλεγα που για, ένα τέτοιο πρόγραμμα έχουμε ένα πλήρες δίκτυο desk ε, για όλες τις συμμετέχουσε χώρες. Και αυτό με χαρά το βλέπουμε και στα ερωτηματολόγια. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει φιλοδοξία και ενθουσιασμός για τη δουλειά αυτή, αλλά παραλλήλως πρέπει να δούμε και τις, ε, τα όρια τις δράσεις των desk αυτών, ε, εις ό,τι αφορά στη νομική βάση του προγράμματος, δεν μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη απόφασης δηλαδή. Ε, χρηματοδοτούνται κατά 50% από την Creative Europe, το άλλο 50% έρχεται από τα κράτη-μέλη και έχουν ενσωματωθεί στην διοικητική δομή των κρατών μελών. Βρίσκονται εκεί προκειμένου να μας βοηθήσουν να εξηγούμε το πρόγραμμα, να εξηγούμε στους ενδιαφερόμενους ε, τις διαδικασίες ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα και υψηλής ποιότητας. Μας βοηθούν και με θέματα διάχυσης και προώθησης. Δεν μπορούν όμως να συμμετάσχουν, να συμμετέχουν στην διαδικασία λήψη απόφασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, είναι πολύ κρίσιμη η χρονική στιγμή σχετικά με την αξιολόγηση των διάμεσων αποτελεσμάτων και των δικτών οι δείκτες είναι ενσωματωμένοι στην νομική βάση του κανονισμού και του προγράμματος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι καθώς εξελίσσεται το πρόγραμμα με την μεταβαλλόμενη κατάσταση που έχουμε μέσα στα χρόνια, οι δείκτες αυτοί ενδεχομένως να μην έχουν παρακολουθήσει με τον καλύτερο τρόπο ε, τις κινήσεις που έχει πραγματοποιήσει το πρόγραμμα. Στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης λοιπόν ε, έχουμε προχωρήσει και σε μια αν θέλετε επανεξέταση των δικτών αυτών και αυτή είναι η στιγμή που θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα των προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί υπό τη Δημιουργική Ευρώπη. Η ε, πραγματική περίοδος επιτήρησης ξεκινάει το 2017 και από εκεί θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την επιτήρηση αυτή με ένα σετ δικτών που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις προτεραιότητες του προγραμμάτου έτσι όπως έχει εξελιχθεί και τροποποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, επίσης έγινε μια ερώτηση σχετικά με το πώς ταιριάζουμε τις υποχρεώσεις προφύλαξης της διαφορετικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Αλλά εδώ είναι μια από τις βασικές προκλήσεις του προγράμματος. Έτσι όπως το θέλησαν οι συνομοθέτες, εξ αρχής Και αυτό ήταν που προσπαθήσαμε να κάνουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, διότι είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματο, λέει ο μιλητής. Σε αυτά θα μείνω, δεν θα πάω στα πιο πολιτιστικά, θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε, καλώ ήλθατε. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη υπόθηκαν. Απλώς θα συμπληρώσω αυτά που είπε ο συνάδελφος. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω την κατάσταση σχετικά με τους ίσους όρους. Υπάρχει ένα σύστημα θετικών διακρίσεων που ε, θεσπίστηκε και δίνει αυτόματα points σε χώρες ε, που, πόντους δηλαδή σε χώρες που έχουν χαμηλή, χαμηλές ικανότητες. Αυτό βασίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού για τη Δημιουργική Ευρώπη που διασφαλίζει ίσους όρους. Ε, προσπαθήσαμε λοιπόν αυτό να περάσει μέσα από τους πόντους. Αυτό το σύστημα, το points system, έχει ελεχθεί, έχει ε, σχεδιαστεί σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη από την Κομισιόν και έχει οδηγήσει, ε, βέβαια μη θελημένα, σε κάποια ε, προβλήματα τα οποία ε, θέλουμε να διορθώσουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασίας ε, της Επιτροπής Προγράμματος του Creative Europe που έχει ήδη συναντηθεί μια φορά και θα συναντηθεί όσες φορές χρειάζεται ώστε να συμφωνήσουμε μέχρι τα τέλη του έτους, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να διορθώσουμε τα προβλήματα και το πρόγραμμα για το 2018 και το πρόγραμμα Creative Europe που θα ξεκινήσει του χρόνου να αντικατοπτρίζουν αυτές τις αλλαγές. Με χαρά θα σας παρουσιάσουμε και τα αποτελέσματα αυτής της ομάδας για τη διευκόλυνση εγγύσεων. Ε, νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε με καθυστέρηση όπως ήδη ε, ε, αναφέρθηκε. Όμως αυτό ε, δεν είναι αλήθεια. Το 2016 ε, στην ουσία ήταν διαθέσιμη, διότι υπήρχε έλλειψη πόρων μέσα στα πλαίσια του του MFF, του Μεσοπρόθεσμου. Ε, γι' αυτό, επειδή ήταν διαθέσιμα τα χρήματα τόσο αργά, η Συμφωνία Ανάθεσης έγινε μέσα, στα, μέσα του έτους και μέχρι τα τέλη του έτους θα μπορέσουμε να υπογράψουμε με τους ενδιαφερόμενους. Όπως καταλαβαίνετε, ε, σε σχέση ε, με ε, άλλα εργαλεία της Κομισιόν, αυτό το εργαλείο, επειδή υπήρχε έλλειψη πόρων, μας επέτρεψε να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε το πεδίο καλύτερα με τους ενδιαφερόμενους, να έρθουμε σε επαφή με τους ενδιαφέρονους του Creative Europe και να μπορέσουμε να κάνουμε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ, ε, Field Forum, ε, συγκεκριμένα θα έχουμε σε 10 μέρη της Ευρώπης και υπήρξε πολύ σημαντική πληροφόρηση μέσω αυτών των ε, εκδηλώσεων προς τον οργανισμό μας. Ευχαριστούμε για τις αυτή αυτές ο ε, του οργανισμού. Ευχαριστώ, είμαι ο Μπράιν Χόλμς, είμαι ο Διευθυντής του Οργανισμού. Σημειώνουμε τα σχόλια για μεγαλύτερη διάδοση των επιτυχημένων ιστοριών και θα δούμε σε συνεργασία με την Κομισιόν πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες ε, για τις επιπτώσεις τώρα. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, Μπορεί να υπάρχουν ε, συγκρούσεις συμφερόντων όταν μιλάμε για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την υποστήριξη των ετούντων. Ε, όμως, ε, για την ε, ε, διοχέτευση των πληροφοριών να πω ότι χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα ερωτηματολόγια, το feedback ε, από τα media desks για να δούμε ποιες είναι οι ανησυχίες τους, για να μπορέσουμε έτσι να πλουστεύσουμε τη διαδικασία και να κάνουμε την κατάσταση πιο ξεκάθαρη για τους ετούντες. Είναι κάτι που ήδη κάνουμε ε, και έχουμε και κάποιες συναντήσεις με τα desks για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα. Όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία, την έχουμε επιταχύνει. Έχει πάει από τους 4,2 μήνες Στου ε, στους 3,96. Και να σας θυμίσω ότι ο στόχος του κανονισμού ήταν 6 μήνες, άρα τα πάμε καλά. Επίσης, αυξήθηκε το επίπεδο feedback που δόθηκε στους ετούντες μέσα ε, από τα, στα πλαίσια του προγράμματος Media για να κατανοούν καλύτερα γιατί υποστηρίξαμε και τους ζητήσαμε να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα desks, ε, να συζητούν γιατί Φυσικά δεν υπάρχει θέμα προστασίας δεδομένων. Ό,τι δίνεται ως πληροφορία πρέπει να γίνεται με τη συνένεση των ετούντων. Τώρα, ε, για να μπορούν οι συνάδελφοι από την Κομισιόν να έχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ των μεγάλων και των μικρών project, να πω ότι τα μεγάλα project είναι η κρίσιμη μάσα, όμως ε, τα μικρά project είναι αυτά που φτάνουν και στους ε, πιο απλούς ανθρώπους στις χώρες. Για το οργανόγραμμα της Κομισιόν και την έλλειψη προσωπικών επαφών προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στο κενό που υπάρχει για τις απαντήσεις στις διάφορες ερωτήσεις. Θέλουμε κάθε φορά οι απαντήσεις που δίνονται να είναι σωστές και χρησιμοποιούμε το σύστημα NING. Ε, είναι σημαντικό βέβαια να γνωρίζουμε σε ποιον μιλάμε και ε, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση για τους ανθρώπους που ε, μπλέκονται όταν απαντάμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για πολύ σύντομη απάντηση θα δώσω στου εμπειρογνώμονε το λόγο γιατί είχαμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η κυρία Λάζαρο, παρακαλώ. Thank you. Ε, ευχαριστώ. από τη δική μου προοπτική κάποιες απαντήσεις όπως επίσης και από την προοπτική του υποπρογράμματος πολιτισμού δεν είναι ακριβώς δύο πράγματα, γιατί είχαμε διαφορετικές απαντήσεις σε μεγάλο βαθμό. Και η προοπτική των εθνικών γραφείων, ε, ανάλογα με το πρόγραμμα που να διαφέρει. Η δημιουργικότητα, ναι, είναι σημαντική. Μπορεί να υπάρχει δημιουργικότητα ως προς την ε, αναδιατύπωση κάποιων συνδυασμών. Γιατί όχι, για να βελτιωθεί παραδείγματι υποστήριξη σε κάποιους τομείς. Πολυγλωσία που αναφέρθηκε, πολιτιστική κληρονομιά. Δημιουργικότητα μπορεί να είναι και ένας τρόπος να ανανεωθούν αυτοί οι τομείς που μπορεί να είναι παλαιοί αλλά και πάρα πολύ σημαντικοί και θεμελιώδεις στην Ευρώπη. Για τις συστάσεις. Είναι οι δικές μου ε, συστάσεις αυτές που σας παρουσίασα σε σχέση με, τις, ε, με την ποιοτική ανάλυση, τις πληροφορίες, που μας έδωσαν τα γραφεία. Και βεβαίω και η επικοινωνία έχει πολύ μεγάλη σημασία και εμεί στο Πανεπιστήμιο μα ιδιαίτερα ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Πρέπει να γίνεται η διάδοση των δεδομένων. Και θα έχει ενδιαφέρον να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Και ανταλλαγή ε, απόρριτων στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καλύτερη ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να ακούσουμε και εσάς να ολοκληρώσουμε. Ναι, πολύ σύντομα για τους δείκτες. που αποτελούν μια καταπροσέγγιση καταγραφή μιας πιο περιπλοκής πραγματικότητας, πιστεύω. Αυτή η καταπροσέγγιση, καταγραφή μας επιτρέπει κάπως να πλωστεύουμε μια κατάσταση, η οποία όμως είναι αρκετά περίπλοκη και δεν μπορούμε να την αναλύσουμε όλοι εδώ. Το σύστημα των δικτών, το πρόγραμμα και ο κανονισμός που έχει εγκριθεί έχουν, πιστεύουμε, επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή το, η διάσταση του Creative Europe μπήκε πολύ αργά στη συζήτηση μέσα από το πρόγραμμα και έτσι για να δώσω και μια θετική εικόνα το σύστημα δεν είναι μόνο να έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα αλλά και να εξασφαλίσουμε τον τρόπο για την καλύτερη κατανόηση του πραγματικού στόχου. Και πρέπει και καλύτερα να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες των δικαιούχων, στους οποίους, τους οποίους προσπαθούμε να πλησιάσουμε και και σε αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο, ιδιαίτερη σημασία να προβάλλουμε τα εθνικά γραφεία να στηριχθούμε στη δική τους δουλειά, όπως είπε και ο κύριος Μόργαν, ώστε να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα συντονισμό, αλλά πάνω απ' όλα να ενστερνίζονται τα προγράμματα. Να κλείσουμε με τον κύριο Μοντό, λοιπόν, τώρα. Α, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ε, πάντοτε ο βασικός δείκτη επιτυχία του προγραμματό είναι ο αριθμό των συμμετοχών. Όσε περισσότερε είχαμε, τόσο μεγαλύτερη απόδειξη θεωρούσαμε ότι είχαμε ότι αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί καλά. Αλλά εκεί είχαμε και κάποιε επιπτώσει τρεβλωτικέ. Γιατί αυτό ο πληθυσμό των συμμετοχών μέσα στον ίδιο φάκελο δημιουργούσε πιέσει, αν θέλετε, συνοστισμό. Για τον αυτοματισμό του προγράμματο αυτό μπορεί να έχει κάποια πλεονεκτήματα και το σύστημα των μικρών, μεσαίων και μεγάλων χωρών ε, η πραγματικότητα παρατηρούμε είναι ότι σε πολλές από τις χώρες Ευρώπης που λειτουργούν τα πράγματα αυτά υπάρχουν διάφορα συστήματα επάλληλα, συμπληρωματικά, περιφερειακά, αναπόλη, με πιστώσεις, με ε, ταμεία υπάρχουν 297 διαφορετικά ταμεία στις διάφορες χώρες. Και σε όλα αυτά οι επαγγελματίες μπορούν να, να στραφούν για ενίσχυση. Έχουμε χώρες που τις θεωρούμε μικρές για την παραγωγή, ως προς την παραγωγή όπως το Λουξεμβούργο, αλλά οι οποίες όπως και η Δανία και η Σουηδία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν διάφορα ταμεία και συστήματα επαγγελματιών. Και γι' αυτό πάμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, το οποίο καθίζεται πιο δύσκολο αν θέλουμε να έχουμε ένα δίκτυ, ένα σύστημα αξιολόγησης, βαθμολόγησης. Και το τελευταίο που μου φάνηκε ε, σημαντικό, ο τομέα εξελίσσεται και εξελίχθηκε. Όλα αυτά που αφορούν στην διάχυση του ψηφιακού υλικού ή του οπτικοακουστικού υλικού, γιατί το πρόγραμμα των media ε, θα μπορούσε να θεωρήσει κανεί ότι ένα πρόγραμμα για τον κινηματογράφο. Αν δούμε όμως το, το Amazon, τη Netflix, όλε αυτέ όλες αυτές εταιρείε βασίζουν την επιτυχία τους ε, σε, τηλεοπτικά serial. Και ξεχνούμε στα πλαίσια του προγραμματό ότι η τηλεόραση σήμερα είναι ε, ένα από, τους, από τις πιο σημαντικέ διόδου διάχυση αυτού του υλικού. Σα ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, για αυτή την παρατήρηση όλες οι μελέτες αυτές που παρουσιάσατε θα είναι μεγάλο ενδιαφέροντος και για εμένα και για τους σκιώδεις και τα υπόλοιπα μέλη αλλά νομίζω και για την Επιτροπή συνολικά. Είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο κάνει εδώ, προχωρεί σε μια έκθεση εφαρμογής και χρειαζόμασταν μια ε, φωνές με κύρος, παρουσιάσεις ε, ερευνητέ με κύρος ε, για να μας βοηθήσει σε αυτήν την διάμεση αξιολόγηση να ευχαριστήσω και την Κομισιόν και τον οργανισμό για την παρουσία της εδώ. Έχουμε, δεν έχουμε πλέον χώρο, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Θα πω απλώς ότι εγώ εκτίμησα το γεγονός ότι υπήρξε μια πολύ ειλικρινής και ανοιχτή ανταλλαγή, αλλά και σοβαρή και το θέμα που δικαίως εδέθη σχετικά με την ένταξη η Επιτροπή ήθελε ένα merging program, ενώ το Κοινοβούλιο θέλησε να αφήσει μια, αν θέλετε, ε, αναγνωρισιμότητα των διαφορετικών σημάτων και λόγο. Ε, υπάρχουν τα διατομικά στοιχεία και τα πολιτισμικά στοιχεία για τα οποία συζητήσαμε την προηγουμένη φορά ότι ήταν το στίχημα της καλύτερης ε, ένταξης. Τώρα με τις δύο γενικές διευθύνσεις και τους δύο επιτρόπους η Κομισιόν πήγε προς μια διαφορετική κατεύθυνση από την ενσωμάτωση αν θέλετε και νομίζω ότι πρέπει να καταβάλουμε κοινή προσπάθεια για να συνδυάσουμε τα πράγματα. Έχουμε μια πολιτική πραγματικότητα που την αναγνωρίζω. Η γάμα δελτα connect και το λέω ξεκάθαρα είναι πολύ πιο προσεκτική σε θέματα copyright, δημιουργών κτλ. Από ό,τι θα ήταν αν δεν είχαμε αυτόν τον διάλογο. Το λέω έξω από τα δόντια. Από, την άλλη μεριά δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από τα χτυλό μας. Το θέμα της διαχείριση και του management υπάρχει. Το θέμα της αυτόματης βαθμολογίας ε, ήταν ε, σημαντικό και μας βοήθησε η προηγούμενη ανταλλαγή που έχουμε και εδώ χρειαζόμαστε συνεργασία με τις ε, κυβερνήσεις και δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνιστικότητας αν μου επιτρέπετε αλλά είναι ενίσχυσης της όλης καλλιτεχνικής και πολιτισμικής παραγωγής. Για, την, για τον οργανισμό υπάρχει ένα θέμα διαφάνειας διαχείρισης. Εγώ είμαι αντίθετη όπως γνωρίζετε με το σύστημα αξιολόγησης που είχε εισαχθεί. Νομίζω ότι και εδώ χρειαζόμαστε κάποια προσπάθεια. Από, την άλλη πλευρά, όπως είπατε σωστά, η νομική βάση δεν αναγνωρίζει συμμετοχή στην διαδικασία λήψη απόφασης στα desk είναι τα κράτη που είναι υπεύθυνα, αλλά εδώ ζητούμε μια συμμετοχή, υπεύθυνη συμμετοχή και συνυπευθυνότητα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ε, μεγαλύτερη συνεργεία και να έχουμε και πιο αντικειμενικές και ανώνυμες εκθέσεις ε, για να κάνουμε την καλύτερη επιλογή. Και το άλλο κεντρικό θέμα που έθεσαν διάφοροι συνάδελφοι είναι η ανησυχία όχι μόνο σχετικά με τα μικρής κλίμακας ε, πρόγραμμα, γιατί έχουμε και ένα δίκτυο στη διαθεσή μας, αλλά και της αίσθηση ότι συχνά δεν μπορούμε να συνδυάσουμε το νόημα της λέξης καινοτομία με την πολιτιστική κληρονομιά και την καλλιτεχνική δημιουργικότητα. πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα αυτά και να μην απορρίπτουμε ή να αποκλείουμε κάτι. Ήδη πολλά είπα, αλλά ήθελα να ε, σημειώσουμε, καθότι το είχαμε συζητήσει και στις 14 Ιουλίου, αλλά θέλαμε να εμβαθύνουμε και με την δική σας συμμετοχή. Τώρα όμως πρέπει να περάσουμε αμέσως σε ένα άλλο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Στο επόμενο σημείο τώρα της μυστικής διατάξεως πάμε την ε, παρουσίαση ε, της κυρίας ε, Χιμένεθ Μπαρμπάτ που είναι εδώ για ανταλλαγή ενημέρωση σχετικά με το έκθεση εφαρμογή για το πρόγραμμα Ευρώπη για του πολίτε. Εδώ έχουμε ε, παρουσιάσει και από το Τμήμα Πολιτικής Β και την Υπηρεσία κοινοβουλευτική έρευνα. Ελπίζω να παραμείνουν συνάδελφοι γιατί είναι σημαντικό ε, να εξετάσουμε δελεχώς ε, ισότιμα όλα τα προγράμματα και έτσι με τη σημερινή συνεδρίαση θα έχουμε ολοκληρώσει την παρουσίαση της, της συζήτησης για τα πιο σημαντικά πολιετή προγράμματα. Τώρα, να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια και μετά οι δύο εμπειρογνώμονες θα μιλήσουν. Παρακαλώ, κυρία Χιμένη Presidenta. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ είμαι η για την έκθεση εφαρμογή για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες που προωθεί το διάλογο μεταξύ των ε, θεσμών της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών. Ή στα πλαίσια του πολιετούς 14-20 ε, προσφέρει οικονομική ενίσχυση για διάφορα προγράμματα για την αδερφοποίηση των πόλεων, μεταξύ άλλων προγραμμάτων για να συνδεθούμε με την ε, συλλογική ευρωακή μνήμη και εδώ προσπαθούμε να υπογραμμίσουμε ε, το ρόλο του Ευρωπαίου πολίτη ως κοινή δίωδο ε, ενσωμάτωσης και ένταξης από διαφορετικές προελεύσεις και πορείες. Και μέσα σε ένα κύμα σκεπτικισμού ε, και περίεργων πολιτικών ισορροπιών θα πρέπει να ενισχύσουμε ακριβώς τη δέσμευση αυτή με τους πολίτες και να πείσουμε, να φέρουμε πίσω κοντά μας, δηλαδή τους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί λόγω έλλειψη εμπιστοσύνη. Και χρειαζόμαστε μετά παραδείγματα για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Θα σας δώσω τρία. Μεταξύ των οργανώσεων που χρηματοδοτούμε είναι το Καφέ Βαμπέλ, που είναι online περιοδικό με ανάλυση σε έξι ευρωακές γλώσσες που το διαχειρίζονται απολύτως ε, σπουδαστές εράσμους. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα πειραματικά προγράμματα συμμετοχής δημοσιογραφίας ε, που τρέχει εδώ και πολλά χρόνια με πρωτοβουλία ακριβώς μικρής ομάδας εφητητών, σπουδαστών που συναντήθηκαν στο Στρασβούργο ε, στα πλαίσια του Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Άλλο ένα παράδειγμα που έχει επιτύχει χρηματοδότηση. European Grassroots Anti-Racist Movement είναι ένα δίκτυο ανθρωπίνων δικαιωμάτων από 33 διαφορετικές χώρες με πρωτοβουλίε δημιουργία ε, κοινωνία των πολιτών ε, για να καταπολεμηθεί η ξενοφοβία, ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός και η άρνηση της γενοκτονίας. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, ε, από την Βαλέθια από το 2015 είχαμε ένα πρόγραμμα για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην Ευρώπη μέσω αδελφοποίησης ευρωπαϊκών πόλεων. Με 8 κοινότητες σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Βέλγιο, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Για να καταλάβετε ότι όταν διαβάζουμε στην πινακίδα η πόλη μας είναι αδελφοποιημένη με την ΤΑΔΕ, πίσω από αυτό υπάρχει μια σημαντική δραστηριότητα και προγράμματα. Αυτά αυτούς τους τελευταίους μήνες είχαμε την ε, ε, δυνατότητα να σημειώσουμε ε, διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν με τους συμμετέχοντες και στην Βαρκελόνη είχαμε πολύ σημαντική συνάντηση ευρωπαϊκοί, ευρωπαίοι πολίτες, κοινωνία των πολιτών σε στιγμές μεγάλων προκλήσεων. Πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε μια, ε, επιτύχαμε μάλλον μια σημαντική εφαρμοσιμότητα του προγράμματος και να ευχαριστήσω τους εμπρεγνώμονες που θα παρουσιάσουν από το, το Ήπειρα ε, και το Τμήμα Πολιτικής Β για κάποιες ιδέες που θα θέλουμε να αναπτύξουμε μέσω της εφαρμογής του προγράμματος αυτού. Καταρχάς θα θέλαμε να, να υποβάλουμε κάποιες συστάσεις σχετικά με τον εξυγχρονισμό της ε, στρατηγικής επικοινωνίας γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα να γίνει πιο γνωστό στην Ευρώπη. Πολλοί πολίτε δεν το γνωρίζουν και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα, κοινων... τα δίκτυα, ε, τα μέσα κοινωνική δικτύωση ε, μέσω έργων και προγραμμάτων που ήδη φίστανται. Όπως το New Narrative for Europe, μεταξύ άλλων. Θα θέλουμε να εμπλωτίσουμε το πρόγραμμα αυτό ε, με στοιχεία που αφορούν τις σημερινές προκλήσεις, να υποστηρίξουμε τη δημοκρατική συμμετοχή μέσω του e-democracy με τους πολίτες, την αδελφοποίηση και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων όπως και πόλεων σε όλο τον κόσμο για ανταλλαγές πολιτισμικές, κοινωνικές και οικονομικές. Και έχουμε και τα προγράμματα της European Remembrance, ώστε η ευρωπαϊκή μνήμη να προασπίσει τις ε, αξίες μας του κοσμικού κράτους που μας ε, έδωσαν ευημερία και ειρήνη. Και για να πάω στο πιο ευαίσθητο θέμα, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 14-20 αφορά συνολικά σχεδόν σε 185 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σημαντικότατη μείωση 13,75% σχετικά με την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο. Εμείς ζητούμε μια ενίσχυση προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να επιβραβεύσουμε τα πιο σημαντικά έργα. Και είναι πολύ περιορισμένο αυτό ο προπολογισμό, ιδιαίτερα να το συγκρίνουμε με τη δημιουργική Ευρώμη και το Erasmus Plus. Εκτιμάται ότι σε, αυτούς, σε αυτά τα δύο πρώτα χρόνια το πρόγραμμα έχει αγγίξει ένα εκατομμύριο πολίτε. Ένα εκατομμύριο Ευρωπαίου πολίτε. Στην περίοδο 7-13 είχαμε εμπλέξει 7 εκατομμύρια Ευρωπαίου πολίτε. Αυτό είναι τεράστιο πλούτο για όλου μα. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ευρωπαϊκές αξίες ένταξης και ενσωμάτωση ενό κοινού προγράμματο μα οδήγησε σε αυτή την περίοδο ευημερία, ειρήνη και ασφάλεια που γνωρίζουμε. Οι αξίε αυτέ ε, μιλούμε σε πάρα πολλά φόρα που ε, τοποθετούνται υπέρ της Ευρώπης, αλλά χρειαζόμαστε μια πραγματική υποστήριξη και χωρί υποστήριξη και ενίσχυση για τα υλικά μέσα και την υποδομή θα είναι απλώς ε, κενά λόγια όλα αυτά. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε μπλοκαρισμένοι, χρειαζόμαστε προσέγγιση με τις, με προς τους πολίτες και τις ενώσεις τους για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές στην απτή πραγματικότητα. Πρόκειται για το μόνο πρόγραμμα που πραγματικά απευθύνεται άμεσα στους πολίτες. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη χρηματοδοτική προσπάθεια και ελπίζω να έχω την υποστήριξη όλων σας, συναδελφοί, για να μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τον προπολογισμό που έχει υποβληθεί. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει η πρόεδρο για αυτήν την εξαιρετική εισαγωγή. Να θυμίσω ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχουμε το σχέδιο έκθεσης και μετά 5 Δεκεμβρίου η συμφορία στην Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Καταρχάς από το EPRS η κυρία Άιζελε. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, για την πρόσκληση να σας μιλήσω και να σας παρουσιάσω σήμερα τα κύρια ευρήματα της έκθεσης μου για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020. Έρχομαι με χαρά να σας μιλήσω. Είναι σημαντικό πιστεύω να μοιραστούμε αυτά τα ευρήματα. Μίλησα νωρίτερα στην αλφή για το EPRS, την αποστολή μας και η έκθεση μου επί, το... επί την ουσία θα είναι πιστεύω χρήσιμη για τη δουλειά σας στην Επιτροπή αυτή. Πρόκειται για έκθεση που ετοίμασα τους τελευταίους μήνες. Καταγράφουμε τα σημεία, τα σημαντικά και τις αδυναμίες των νέων δομών καταγράφουμε κάποια πρώτα ευρήματα και συστάσεις και ξεκινώ επισημένως το πρόγραμμα υπάρχει μόνο δύο χρόνια τώρα δεν είναι πολύ ο χρόνος πρέπει να έχουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο εφαρμογής Σύντομα τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο πρόγραμμα, στο προηγούμενο δηλαδή πρόγραμμα, και να υπογραμμίσω τις δυσκολίες του, τις ελλείψεις του. Όπως αυτές καταγράφηκαν το Σεπτέμβριο 2015 στην Εξπόσταση Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το προηγούμενο πρόγραμμα είχε αξιολογηθεί θετικά, κρίθηκε επιτυχημένο. θεωρήθηκε ότι διαφοροποιείται αρκετά σε σχέση με το πεδίο του, του στόχους του, τα, το αντικείμενό του από άλλα προγράμματα. Προσθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταγράφεται ότι μπορεί να καταστήσει δυνατές δραστηριότητες που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν το πρόγραμμα αυτό. Και επίσης με την αξιολόγηση αναφέρεται ότι δραστηριότητες ε, μετά την ολοκλήρωση των έργων και παρακολούθηση έχουν πολύ μεγάλη σημασία για να υπάρχουν απτά αποτελέσματα. Εάν δεν υπήρχε δηλαδή επαρκές ε, και αξιόπιστο follow-up, δεν ήταν ορατά τα αποτελέσματα. Επίσης και εν τέλει καταγράφουμε ότι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος μπορεί να ενισχυθεί εάν δοθεί περισσότερη έμφαση σε έργα που θα έχουν τον ε, πολίτη στο πιδάλιο. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί πρόκειται για το μόνο πρόγραμμα που απευθύνεται απευθείας στον πολίτη. Θα ήθελα επίσης να παρουσιάσω κάποια προκαταρκτικά εύρηματα της δικής μου έκθεσης. Ανέφερα προς βρισκόμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο. Προβλέπουμε τη συνέχιση της επιτυχίας των προηγούμενων προγραμμάτων στην Ευρώπη και πέραν αυτής. 2.000 οργανώσεις στην Ευρώπη συμμετέχουν απευθείας περί το 1 εκατομμύριο πολιτών έχει άμεση ή έμεση εμπλοκή στα ε, έργα. Η υλοποίηση προχωρεί απρόσκοπτα, η διαχείριση του προγράμματος είναι σταθερή, στα χέρια της ΕΑΣΕΑ και της DG ε, στο Δικαιοσύνης Home ε, που ανέλαβε από την ΚΟΜ πέρσι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετανάστευση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την διαπολιτισμικότητα πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας δηλαδή. Πάντως, και ήδη αναφέρθηκε και νωρίτερα, η χρηματοδότηση και η ορατότητα έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δηλαδή ε, επαρκής εκπροσώπηση έργων μικρού προϋπολογισμού με επαρκείς στόχους και φιλοδοξίες με 250 εκατομμύρια χρηματοδότηση το προηγούμενο πρόγραμμα το τωρινό έχει τώρα 185 εκατομμύρια όπως άλλωστε ακούσαμε και νωρίτερα. Συνεχίζω επίσης λέγοντας ότι ο αριθμός των ε, αιτήσεων που διατυπώνονται υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος και την ανάγκη να δοθεί συνέχεια και να επεκταθεί ενδεχομένω. Είναι ανταγωνιστικό. Είχαμε 280.000 αιτήσει από τις οποίες 400 μόνο εγκρίθηκαν μέσα το 2015 και επίσης από τα όσα μάθαμε με την έρευνα μας ήταν τα έργα ιδιαίτερη ποιότητας και πολλά αξιόλογα ε, έργα προτάσεις έργων χρειάστηκε να απορριφθούν γιατί δεν επαρκούσαν οι δυνατότητες. τις δραστηριότητες για σταθερότητα και ορατότητα, επιλογή έργου εξισορροπημένη και γεωγραφικά. Άλλωστε αυτή ήταν και μια από τις παρατηρήσεις της προηγούμενης αξιολόγησης. Τώρα λοιπόν έχουμε μια καλύτερη γεωγραφική κατανομή. και έχουν συμπεριληφθεί και δείκτες ε, επιδόσεων. Συστάσεις λοιπόν. Πρώτον και σημαντικότερο κύριο μήνυμα ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Σημαντικά προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι του, να, ε, να εξασφαλίζεται η λειτουργία του και η ορθή εφαρμογή του. Δεύτερο, η σύσταση θα πρέπει να ε, γίνεται η κατανομή των πόρων, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό κατά 20% στο πρώτο σκέλος, ευρωπαϊκή μνήμη, 60% στο δεύτερο σκέλος, δημοκρατική συμμετοχή. Η δε έρευνά μου δείχνει ότι το σκέλος υπαριθμών 1 κατά 2014 και 2015 ήταν ε, σε ένα ποσοστό χρηματοδότησης λίγο χαμηλότερο από το 20%, άρα θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη και για το μέλλον του προγράμματος. Και επίσης, εν τέλει, η χρηματοδότηση που προβλέπεται ε, για την Ευρώπη για τους πολίτες θα πρέπει να χορηγείται και να χρησιμοποιείται για τους στόχους του προγράμματος γιατί συχνά πάει, πάνε οι πόροι στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, που βεβαίω έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά είναι άλλη υπόθεση αυτή και άλλο το να περικόπτονται στη συνέχεια κονδύλια τα οποία είχαν χορηγηθεί για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ και σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήσταν πολύ ακριβείς. Μας δώσατε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Και τώρα δίνουμε το λόγο στην κυρία Τζέφρις. Την κυρία Τζέφρις, η οποία θα μας δώσει τα πορίσματα των εργασιών που ανέλαβε από το Τμήμα Μελετών του Κοινοβουλίου, θεματικό ε, σκέλος Β, για τις ε, την υλοποίηση νέων προγραμμάτων, μια μελέτη η οποία στηρίζεται από ό,τι έχω καταλάβει σε συνεντεύξεις και θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα ασφαλώς. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Mm-hmm. Uh, I'd like to... Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον συνάδελφο Bradford, ο οποίος ε, ε, θα κάνει την παρουσίαση. Πρώτος. Όχι, εσείς αρχίζετε. Ωραία. Πολύ καλά. Καλησπέρα. Είμαι ο Bradford Ρόμερ και η Ρίνα Τζέφρις και εγώ δουλεύουμε για μια εταιρεία συμβούλων που ονομάζεται Coffee που είναι μια σειρά κοινωνικών ερευνητών που κάνει ε, έρευνες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Βρετανική Κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις. Θα σας μιλήσουμε εδώ για μια μελέτη που εγώ και η Ρίνα κάναμε για το Europe for Citizens, το πρόγραμμα, δηλαδή η Ευρώπη για τους πολίτες, εγώ είμαι Αμερικανός και μάλλον ο μοναδικός στην αίθουσα που δεν είναι Ευρωπαίος ε, πολίτης. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και πάντοτε έχω την Ειρήνα να με υποστηρίζει. Ο σκοπός ε, της συζήτησης ε, αυτού του, σήμερα είναι να σας παρουσιάσουμε τη μικρή μας μελέτη. Όπως ήδη ανέφερε η συγκήτρια και η πρόεδρος, μιλάμε για ε, κάποιες με εθνικά σημεία επαφής που βοηθούν τους ανθρώπους και τους οργανισμούς να εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Όπως υπόθηκε, αυτό το πρόγραμμα είναι από τα μοναδικά ή ίσως το μοναδικό που στοχεύει στους ίδιους τους πολίτες με τόσο άμεσο τρόπο. Περισσότερο λοιπόν από ότι σε άλλα προγράμματα, τα εθνικά σημεία επαφής παίζουν σημαντικό ρόλο και όπως είπε και η ε, καθηγήτρια κυρία Λατσάρο, στην προηγούμενη παρουσίασή της, ε, τα εθνικά σημεία επαφής είναι σε καλή θέση, δίνουν ε, πολύ πληροφορημένη ε, πολύ καλή περιστατωμένη πληροφόρηση και υπάρχουν εκεί για αρκετό διάστημα. Όπως γνωρίζετε ήδη, το Europe for Citizens είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους που το χρειαζόμαστε αυτό. Οι περισσότεροι από εσάς εδώ το γνωρίζουν καλύτερα από μένα. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν το οποίο ξεκίνησε ξανά το 2014 μέσα στα πλαίσια μιας νέας χρηματοδοτικής περίοδου. Έκτοτε έχει γίνει, μέχρι τότε μάλλον, είχε χάσει την εστίασή του και κάπως κολυσιακούσαν οι διαδικασίες. Το νέο πρόγραμμα λοιπόν προσπαθεί να είναι πιο απλό και πιο στρατηγικό σε επίπεδο στόχων. Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν τρέχει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο διάστημα δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι επαρκές για να ελέγξουμε κάποια στοιχεία από το νέο πρόγραμμα, μιλώντας με τα εθνικά σημεία επαφής τον Απρίλιο και τον Μάιο. Αυτό κάναμε δηλαδή. Κάναμε συνεντεύξεις με 24 σημεία επαφής σε εθνικό επίπεδο και προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες απαντήσεις, κάποιες συστάσεις και να βγάλουμε κάποια σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουμε ζητήματα προπολογισμού και άλλα ζητήματα που είναι δύσκολα να αλλάξουν. Εγώ και η Ειρήνα λοιπόν θα σας μιλήσουμε για τα βασικά βρήματα και τα συμπεράσματα και αυτό ελπίζω να οδηγήσει σε επιπλέον συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μπραντ, λέει η Ειρήνα. Ας, ε, θυμίσω λοιπόν και εγώ τη σημασία αυτή τη ε, ε, μεθόδου. Βασίστηκε σε... Ε, συνεντεύξεις, δεν είναι πλήρης αξιολόγηση, είναι μια ένδειξη όμως ε, των περιοχών ενδιαφέροντος, τι μπορεί να βελτιωθεί, ε, πού υπάρχουν ανησυχίες, ε, τι μπορεί να πάει καλύτερα. Στις επόμενες διαφάνειες λοιπόν έχω συναψίσει τα βασικά ζητήματα και τα έχω ομαδοποιήσει βάσει των βασικών στόχων της ε, έρευνας, ε, δηλαδή ποιες είναι οι, ε, οι διάφορες του προγράμματος, εθνικά σημεία επαφής. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε τα βασικά ευρήματα και να κάνουμε κάποιες συστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια ότι όταν κάναμε τις συστάσεις, σκεφτόμασταν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και δεν αμφισβητούσαμε τη δυναμική βάση του προγράμματος. Ήταν πιο πρακτικές και όχι τόσο ρηξικέλευτες οι προτάσεις. Ε, ας δούμε τώρα ποιες είναι οι βασικές αντιλήψεις των εθνικών ε, σημείων επαφής. Η αναθεώρηση φυσικά βελτίωσε το πρόγραμμα, διότι υπήρξε μια καλύτερη διευθέτηση των δραστηριοτήτων. Και ένα άλλο στοιχείο που τα εθνικά σημεία επαφή καλωσόρισαν ήταν ότι υπήρχε εκ των προτέρων ανακοίνωση των εθνικών προτεραιοτήτων και μπορούσαν να κάνουν αίτηση για πολλά έτη και όχι ε, για ένα έτος μόνο. Άρα είχαν τη δυνατότητα οι ετούντες σε περισσότερο χρόνο να σκεφτούν την αίτησή τους και να την αναπτύξουν. Αυτό φυσικά είχε ως αποτέλεσμα ε, το πρόγραμμα να είναι πιο κατανοητό ε, για τους ετούντες από την πλευρά δηλαδή των εθνικών σημείων επαφής που οδηγεί και σε καλύτερη ποιότητα project. Διότι οι στόχοι είναι πιο κοντά στα θέλω των ετούντων και παράγουν πιο σταθερά και συνεκτικά project. Σκεφτόμενοι λοιπόν τις προτεραιότητες του προγράμματος. Κάποιες θεωρήθηκαν πολύ γενικές ή πολύ επικεντρωμένες στο παρελθόν. Υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία επίσης που αναφέρθηκαν πολύ σημαντικά. Ο οδηγός του προγράμματος για παράδειγμα δεν ήταν ο κατάλληλος ως έχει. Καταλήξαμε λοιπόν σε δύο συστάσεις. Πρώτον, ότι η Κομισιόν θα πρέπει να, να διατυπώσει κάποιες από τις προτεραιότητες του προγράμματος ε, ώστε να συνάδουν με το ε, πλαίσιο των ευρωπαϊκών Ε, Το 20% του ε, προγράμματος του προϋπολογισμού δίνεται στην μνήμη, όμως θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες επιλογές για τους ετούντες σε αυτό το τομέα. Επίσης υπάρχει μεγάλη επικέντρωση στο σταλινισμό και τον εθνικό σοσιαλισμό, κάτι που αποκλείει πολλούς από τη συμμετοχή. Οι στόχοι του προγράμματος επίσης θα μπορούσαν να απλουστευτούν περαιτέρω, όπως έγινε και με την αναθόρυση του 2014, όμως αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς να επαναδιατυπώσουμε και τη νομική βάση. Άρα στο μέλλον θα το δούμε αυτό. Τελεία. Μια πολύ σημαντική αναφορά για τη σημεία επαφής και τους ετούντες είναι ο οδηγός. Αναφέρθηκε σε πολλές συνεντεύξεις που είχαμε με τα εθνικά σημεία επαφής ότι κάποιες φορές αυτός είναι ατελής, περίπλοκος και θα θέλανε περισσότερη καθαρότητα στα κριτήρια επιλογής και τις οικονομικές πτυχές του προγράμματος. Πάμε τώρα στα οικονομικά στοιχεία και τη διαδικασία αίτησης. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το εφάπαξ σύστημα τονίστηκε ως μια βελτίωση, μεγάλη βελτίωση μάλιστα, από την πλευρά, από την, κατά την άποψη των εθνικών σημείων επαφής. Και από την πλευρά των ετούντων. Όμως, όπως έχουν τα πράγματα τώρα, υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποιες ε, λεπτομέρειες στην χρηματοδότηση που είναι ασαφείς και θεωρούνται δυσκολίες. Ας πούμε ότι η προχρηματοδότηση είναι 50% μόνο και υπάρχει μια απέτηση για συγχρηματοδότηση. Κάποιοι οργανισμοί, ειδικότερα μικροί, με λιγότερες οικονομικές δυνατότητες ή που είναι από κράτη-μέλη όπου υπήρξε μια στεναρή οικονομική κρίση, ε, παλεύουν για να αντιμετωπίσουν αυτά τα κριτήρια. Επίσης, οι γεωγραφικές διαφορές ως προς το ε, κόστος διαβίωσης ε, επηρεάζουν τις χορηγήσεις. Ξέρω ότι αυτό γίνεται σε άλλα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Erasmus+. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα ήταν καλό να υπάρχουν γεωγραφικές διαφορές, να υπάρξει μια αναθεώρηση σε αυτό το κομμάτι. Γενικά η διαδικασία αίτηση είχε καλή και θετική αξιολόγηση από τους ετούντες, σύμφωνα με τα εθνικά σημεία επαφής, κυρίως λόγω της ηλεκτρονικής αίτησης παρόλο που υπήρξαν κάποιες μικρές δυσκολίες που αναφέρθηκαν, όμως ένα θέμα ε, που τέθηκε ήταν ο τρόπος που δίνεται πληροφόρηση σε όσους απορρίπτονται. Ίσως ε, να γίνει κάτι διαφορετικό. Τώρα υπάρχει μια επιστολή στάνταρ, επιστολή τυποποιημένη, που απλώς λέει ότι Εντάξει, ε, απορριφθήκατε, δεν δίνει περισσότερους λόγους, οπότε οι ετούντες χάνουν την ευκαιρία να μάθουν πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη θέση τους σε, μια δεύτερη, ε, σε ένα δεύτερο διαγωνισμό, σε μια δεύτερη προκήρυξη. Τώρα υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των ε, φιλόδοξων στόχων του προγράμματος και των ελάχιστων χρηματοδοτικών ευκαιριών. Πώς το αντιμετωπίζουμε θα μπορούσαμε να συστήσουμε αύξηση του προπολογισμού που θα ήταν το πιο σημαντικό φυσικά, όμως παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και κάποια από τα modules χρηματοδότησης. Επίσης, μπορούμε να βελτιώσουμε και τον τρόπο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Ας πούμε, τα εθνικά σημεία επαφής θα μπορούσαν να έχουν μια πιο επίσημη θέση. Η επικοινωνία λοιπόν γενικά φαίνεται ότι ήταν ε, ε, ικανοποιητική παρόλο που τα εργαλεία θα μπορούσαν να βελτιωθούν ειδικότερα όσον αφορά το πόρταλ των επιτυχημένων project που είναι μια καλή ευκαιρία αλλά θα μπορούσε να βελτιωθεί και η ιστοσελίδα θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστική και πιο, ε, να προσφέρει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. Επίσης γενικά φαίνεται ότι ε, από το 2014 στο 2015 είχαμε ε, σε πάνω από 2.000 project ε, χρήση αυτών των εργαλείων, άρα θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το επίπεδο ευαισθητοποίησης των ομάδων που στις οποίες στοχεύουμε οι οποίες έχουν αυξηθεί από το 2014. Τώρα για τα σημεία επαφή, να πω ότι γενικά είναι ικανοποιημένα με τη θέση τους, όμως υπάρχουν κάποιες δυνατότητες να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό τους. Ας πούμε, όπως γίνεται με τα Creative Europe Desks, θέλουν και αυτά να είναι περισσότερο στα πράγματα να εμπλέκονται περισσότερο, να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες από την Επιτροπή Προγράμματος και οι απόψεις τους και η εμπειρία τους θα ήταν καλή κατά την ε, αναθεώρηση και αναδιατύπωση του οδηγού. Γιατί έχουν και επαφή με τους βασικούς εμπλεκόμενους, στη βάση δηλαδή του προγράμματος. Επίσης, η συνέργεια μεταξύ του Europe for Citizens και άλλων προγραμμάτων ε, ή όμοιας φύσης πάντοτε, θα, πάντοτε προσφέρει θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Bene, Σας ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίαση αυτή. Δώσω τώρα το λόγο στους Κιώδης. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις από ό,τι καταλαβαίνω από τον, από τον συνάδελφο Ράιαν και από τον κύριο Γκίου. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Νομίζω ότι πολλά από αυτά που διαπίστωσε η έρευνα ε, ήδη είχαν αναδυθεί στις συζητήσεις μας με τους stakeholders και τους ετούντες ε, ε, στα εθνικά σημεία επαφής τους εθνικούς οργανισμούς. Ε, σήμερα λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από το Σαντιάκο ε, Φίσ, εκ μέρους του Φίσας που δεν μπορεί να έρθει από τη χώρα των Βάσκων να πω ότι το πρόγραμμα Europe for Citizens είναι πολύ σημαντικό και ε, υπό το φως αυτών που συμβαίνουν με το Brexit στην ε, Ηνωμένο Βασίλειο ε, θέλουμε οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αισθάνονται ενωμένοι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες λαϊκιστικές ε, τάσεις και τα κινήματα, να υπάρχει καλύτερη γνώση της Ευρώπης, να μεγαλώνουμε και να προοδεύουμε όλοι μαζί. Αυτά να περνάνε και λυπόμαστε που ακριβώς σε αυτόν τον τομέα, στα κράτη-μέλη, έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός ε, και προτείνονται και άλλες ε, μειώσεις από την Κομισιόν. Ε, βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι εμείς ως Κοινοβούλιο να μαχηθούμε ώστε ε, αυτό το πρόγραμμα να έχει τα κατάλληλα ε, χρηματοδοτικά μέσα. Επίσης, καταλαβαίνουμε από όσα παρουσιάσατε ότι είχαμε καλά προγράμματα, πολύ ε, καλά προγράμματα και αυτοί που έκαναν τις αιτήσει ε, δεν κατανοούσαν γιατί απορρίφθηκαν πολλές φορές. Εμείς ε, λένε πληρούμε τα κριτήρια. Έχουμε προγράμματα τα οποία προέρχονται από πολίτες και όχι από οργανισμούς. Και υπάρχει μεγάλη ποικιλία, παρόλα αυτά υπήρξε απόρριψη και δεν γνωρίζουν για ποιο λόγο. Σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν είμαστε αντιπαραγωγικοί, ιδιαίτερα αντιπαραγωγικοί, γιατί δεν έχουμε και την αιτιολόγηση των απορρίψεων και υπάρχει και μία δυσαρέσκεια εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν μπορεί κανείς να απολαύσει τα προνόμια από αυτά τα προγράμματα. Αυτό να ρωτιέμαι λοιπόν, ε, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Και να ρωτιέμαι λοιπόν, ποια θα είναι η επίπτωση μιας περαιτέρω μείωσης του προϋπολογισμού θα δείξουμε μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Νομίζω ότι πολλοί γνωρίζουν το πρόγραμμα, αλλά δεν θέλουν να συμμετέχουν γιατί πάρα πολλές φορές μπήκαν στον κόπο να κάνουν αίτηση αλλά ε, δεν ε, έγιναν δεκτές οι αιτήσεις λόγω της μεγάλης ε, διοικητικής διαδικασίας. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να μην ε, τοντίζουμε περισσότερο τα κακά από τα καλά, να ε, βελτιώσουμε το πρόγραμμα έτσι ώστε να γίνει πιο κατανοητό στον κόσμο ε, να, και όπως είπατε τα βασικά σημεία του προγράμματος έχουν να κάνουν με, τα, με τους εθνικούς οργανισμούς. Αυτοί πρέπει να τα κατανοούν καλύτερα, να είναι πιο διακριτά σε αυτούς, γιατί όταν υπάρξει αυτή η προϋπόθεση θα είναι πιο εύκολο να Παρέχουμε όλα όσα ε, διατίθενται, ακόμα και το, η δυνατότητα online. Να δούμε ε, πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα, ας πούμε, της αγραμματοσύνης, πράγματα που και αυτά ε, ε, εμποδίζουν τον κόσμο να συμμετέχει. Θα ήταν καλό λοιπόν να, και θα με ενδιέφερε να δω ε, πώς θα μπορούσαμε μέσα από εθελοντικά προγράμματα που προέρχονται από τους ίδιους τους πολίτες να έχουμε περισσότερα project για να μπορέσουμε να τους δώσουμε μια καθοδήγηση μέσα από επαγγελματίε, έτσι ώστε τα μικρά και μεσαία project ε, που είναι από τους πολίτες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τα μεγάλα project διότι ε, και για τις κοινωνικές, ε, κοινωνιολογικές ε, μελέτες θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια επαναχρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ κυρία Αγγιό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Όλα αυτά που θα μας βοηθούσαν να καταπολεμήσουμε το σκεπτικισμό, να κατανοήσουμε καλύτερα τη διαφορετικότητα και τις κοινέ αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την αλληλοκατανόηση, το διάλογο, τον διαπολιτισμικό ε, στην αρχή του δευτέρου αυτού εξαμήνου έχουν ιδιαίτερη σημασία. Και νομίζω ότι είναι σωστό και καλό να μπορούμε ε, να συζητούμε για τέτοια πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν μια ερώτηση διευκρίνησης προς μελετητές ε, και μια-δύο παρατηρήσει που θα μπορούσαν να συμφωνήσουν και με τους συναδέλφου. Καταρχάς το δυναμικό αυτών των σημείων επαφή. οι δυνατότητες που έχουν. Έχετε έρθει σε επαφή με διαφόρους, ε, υπάρχει και μια ετερογένεια ε, της σύνθεσης αυτών των σημείων επαφή. Εσείς θεωρείτε ότι εκεί υπάρχει ένα δυναμικό προς ανάπτυξη. Και γίνεται καλύτερος συντονισμός εδώ. Και για να μείνω εντός του χρονικού πλαισίου που έχω, θα μπορούσε να σημειώσει κανείς ε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της νομικής ε, βάσης του προγραμματός ε, έχει περιορισμένε αρμοδιότητες κυρίως συμβουλευτικέ. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς για το μέλλον, ενδεχομένως να έχουμε έναν πιο ενισχυμένο ρόλο στα πλαίσια ενό τέτοιου προγράμματος για τη χρηματοδότηση τι θα επανέλθω, νομίζω ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά προς τα οποία συμφωνώ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διαρευνηθεί κάθε δυνατότητα ενίσχυσης, αύξησης, εντός των προτεραιοτήτων θα μπορούσαν να επανεξεταστούν και ακόμα περισσότερο όπως και αυτό ελεγχθεί, καθότι έχουμε διαφορετικής κλίμακας προγράμματα. Τα λεγόμενα μικρά δεν είναι αναγκαστικά δεν τα χαρακτηρίζουμε έτσι για να τα επικρίνουμε. Χρειαζόμαστε καλύτερη δημοσιονομική αποτελεσματικότητα και χρειαζόμαστε και δυνατότητα ανάπτυξη και μικρότερη κλίμακα προγραμμάτων. Τώρα βεβαίω ε, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία η περιπλοκότητα της κατάστασης είναι γνωστή και δύο τελευταία σημεία αναφέρθηκα στο συντονισμό μεταξύ των σημείων επαφής με την ετερογένεια που έχουν Άρα το τελευταίο σημείο που έχω είναι το θέμα της επικοινωνίας. Είμαστε στην ψηφιακή εποχή, έχουμε κοινωνική δικτύωση. Εγώ και λόγω ηλικίας δεν έχω ενδεχομένως απόλυτος πλήρη εικόνα ε, της ανάπτυξης όλων αυτών και ιδιαίτερα ε, των σημείων επαφή, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο διαδραστικά, πολύ πιο παρόντα στο διαδίκτυο με ένα λόγο και μια τοποθέτηση λιγότερο γραφειοκρατική και πιο παιδαγωγική. Αυτές θα ήταν οι παρατηρήσει μου και οι προτάσει μου αν θέλετε. Ευχαριστούμε Σιλβί. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να ακούσουμε και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που την ευχαριστώ για την συμμετοχή. Α, έχουμε ακόμα μία συνάδελφο που ζήτησε το λόγο. Δεν, δεν σας είχα δει, ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ έκανα μία πρώτη μελέτη της παρουσίασης των μελητών και έχω ήπιες απορίες και άκουσα και τις αναφορές του στα εθνικά σημεία επαφής. Οι απορίες μου είναι ακριβώς σχετικά με την σχετική αναλογία που υπάρχει στο πρόγραμμα πέρα από τα μεγέθη που ήδη παρουσιάστηκαν και τα γνωρίζουμε. Αλλά στη δομή του προγράμματο, σε εκείνο το τμήμα, μεταξύ των προτεραιοτήτων, διαβάζει κανεί, όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε το θέμα του ευρωσκεπτικισμού και να το συζητήσουμε. Δηλαδή μιλούμε για την αναγκαιότητα να ε, αναγνωρίσουμε όσο γεγονός το φαινόμενο αυτό, αλλά με ανησυχεί με ανησυχεί και το μέσο μέσο του οποίου θα θέλαμε να δώσουμε απαντήσει, δηλαδή η γραμμή χρηματοδότησης τη Ευρωπαϊκής Συντροπή για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τώρα, ε, αισθάνομαι εδώ μία υποψία υποκρισίας made in Europe. Δεν ξέρω, πολύ αμφιβάλλω θα μπορούσε να συζητηθεί το θέμα του ευρωσκεπτικισμού σε ένα τέτοιο πλάσιο, πλαίσιο με προαποφασισμένες γραμμές δηλαδή από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμπολίτε μου στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια έχουν απομακρυνθεί όλο και περισσότερο. Κοιτούν με καχυποψία και απογοήτευση την Ευρώπη και αυτή αυξάνεται. Και αυτό για διάφορους λόγους. Οικονομικούς, πολιτικούς και λόγου ταυτότητο Αναμφίβολα η οικονομική κρίση έχει ενισχύσει αυτέ τι τάσει. Και σήμερα η πρόκληση είναι η δυνατότητα των θεσμών να αντιμετωπίσουν τα αιτήματα και τις ανάγκες των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πάντα θεωρεί το από σημαντική των πολιτών ως ανίδα σωτηρίας, αλλά δεν είναι πλέον έτσι. Έχουμε έντονο πεσιμισμό και απεσιοδοξία που επικρατεί. Υπάρχει λοιπόν ένα παράδοξο να επενδύουμε τα χρήματα των συμπολιτών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να συζητήσουμε και όχι να αποσιωπήσουμε, ελπίζω, ένα φαινόμενο που είναι πλέον προφανέστατο για όλου. Οι αιτίε είναι προφανεί και δεν πρόκειται να το επιλύσουμε με εκδηλώσει και συναντήσει και μελέτε. Προ Θεού, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για όλου αυτού που δεν έχουν φωνή, αλλά ε, φοβούμαι ότι όλα αυτά μπορεί να αποδειχθούν ε, φούσκα, για να το πω έτσι και στηρίζομαι και σε κάποιε παρατηρήσει των μελετητών, των εμπειρογνωμόνων που υπογραμμίζουν κάποιες, ε, ε, κάποια αδύνατα σημεία. Τη συγχρηματοδότηση, το πόσο είναι δύσκολο σε περίοδους κρίσης όπω σήμερα για αρκετέ χώρε να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα, να διαχειριστούν τέτοια μέσα χρηματοδοτικά. Επίση δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστο ζωή, που είναι πολύ διαφορετικό μεταξύ των διαφόρων χωρών. Και ολοκληρώνω με μια ερώτηση. Ήθελα να κατανοήσω συγκεκριμένα τι εννοεί η εμπειρογνώμων όταν μιλάει για ένα 20% του Strand 1 που είναι στην ουσία λιγότερο από 20% για την περίοδο 14-15. Ίσως μέσω διερμηνίας έχασα κάπως αυτό που λέγατε. Ήθελα να καταλάβω καλύτερα το ποσοστό. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, το λόγο έχει η Κομισιόν και την οποία ευχαριστώ. Head of Unit Institutional Relations της Delta ε, Home. Και ο επικεφαλής ε, κύριος Πιλάγιο. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που ανέλευε αυτή την δραστηριότητα. Πράγματι του χρόνου πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει την αξιολόγηση του προγράμματος και έτσι όλα όσα ακούγονται σήμερα μπορούμε να ε, χρησιμεύσουν και να εμπλουτίσουν τη δική μας αξιολόγηση. Γιατί μια πρώτη λοιπόν εικόνα το 2007-2013 ήταν επιτυχημένο. Πολλά διδάγματα αποκομίσαμε και τα ενσωματώσαμε στο νέο πρόγραμμα, τους καταστήσαμε πιο απλό, άμεσο και έτσι είδαμε αποτελέσματα και ως προς την γεωγραφική κατανομή και ως προς τον αριθμό των αιτήσεων και πολλά άλλα. Βέβαια, βελτίωση πάντα χωρί. Και νομίζω ότι πολλές από τις προτάσεις που ακούστηκαν μπορούν να εξεταστούν με σοβαρότητα και να ενσωματωθούν στα περαιτέρω, στα περαιτέρω προτάσεις μας. Βεβαίως είναι πάντα πηγή δυσφορίας το να απορριφθεί μια αίτηση και εμείς με χαρά βλέπουμε την έγκριση των αιτήσεων που ε, προχωρεί, προχωρούν και πάντα βέβαια υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Νομίζω ότι μπορούμε να επαναλάβουμε τα, τις εμπειρίες των προηγουμένων ετών, να τις αξιολογήσουμε και να, να βελτιώσουμε τα προγράμματα για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία ηγήτρια, κυρίες και κύριοι. Θέλω και εγώ να συνεχίσω με τις, προσ... με τις προτάσεις μας από πλευράς της ε, ε, δικής μας υπηρεσίας για την εμπειρία του 2014-2015. Όντως έχουμε επιτύχει τον επιδιωκόμενο στόχο, το 20% δηλαδή που έπρεπε να ενσωματωθεί και αυτό με τα operating grants μαζί που θα ήταν τα λειτουργικά εκείνα βοηθήματα που ε, καλύπτουν τα έργα μνήμης. Και ίσως αυτό βλέπετε την ε, απόκληση στην ε, ανάλυση. Βεβαίως ε, οι δυνατότητες χρηματοδότησης και το cash flow, η ρευστότητα για την κοινωνία των πολιτών πολλές φορές είναι περιορισμένη και γι' αυτό κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερες ε, διευκολύνσεις πάντα αυτό στο ε, βαθμό που μας το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες του κάθε ετήσιου προϋπολογισμού και αυτό πάντα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Σε σχέση με παρατηρήσεις που ακούστηκαν, τη διατύπωση του προγράμματος, την ανάγκη να αποφεύγεται η ιδιόλεκτος εκείνη η οποία πολλές φορές αποτελεί φραγμό και δεν επιτρέπει την κατανόηση, βεβαίως και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει τις προσπαθίες μας. Είμαστε σε επαφή με, τις, με τους φορείς σε εθνικό επίπεδο και τις επαφές μας, ώστε να καθιστούμε όσο δυνατόν πιο κατανοητά τα κύβερνα που αποστολούμε στους πιθανούς ε, εταίρους και συνεργάτες. Για το feedback και την, ε, τις απαντήσεις εκείνους που δυστυχώς πρέπει να απορρίψουμε και είπατε ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό το ποσοστό επιτυχίας του προγράμματος. Ε, θα κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την επικοινωνία με εκείνους που θα αναγκαστούμε να απορρίπτουμε δεδομένων δε και των πολυάριθμων αιτήσεων και του γραφειοκρατικού κρατικού κόστους που θα ε, σήμαινε η προσωπική διατύπωση της σχετικής επικοινωνίας και η παρακολούθηση της κάθε αιτήσεως σε ατομικό επίπεδο. Η ιδιαιτερότητα του προγράμματο λοιπόν είναι ότι απευθύνεται κυρίω σε οργανώσεις Κοινωνία των πολιτών που δεν καλύπτει άλλο πρόγραμμα τη ε, Ευρωπαϊκής Ένωση, από ό,τι γνωρίζουμε. Ε, είναι μια σημαντική λοιπόν ιδιαιτερότητα και θέλω ιδιαίτερω να σημειώσω ότι ο μέσος όρος των προγραμμάτων και ιδιαίτερα η αδελφοποίηση πόλεων και ακόμα και σε μικρά ε, έργα μέχρι 5.000 ευρώ η παραδείγματη, πολύ μικρή χρηματοδότηση, προσπαθούμε πάντοτε να, κατα, ε, να αγγίζουμε να φτάνουμε μέχρι το χαμηλότερο πιθανό επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών ώστε να τους πλησιάζουμε, ώστε να έχουμε την επαφή μαζί τους. Ε, Επίση θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει μια μορφή ε, επικοινωνίας και προσπαθούμε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τη διαθεσιμότητα της Κομισιόν ε, και για την ε, στήριξη προς τους ε, εισηγητές για την βοήθειά σας. Αν θέλετε να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις που ετέθησαν και μετά θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να κλείσει. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποιες απαντήσεις στα σχόλια που έγιναν από, το, κίν τους Ευρωβουλευτές όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του προγράμματος Europe for Citizens και του ευρωσκεπτικισμού. Να πω ότι είναι αλήθεια πως είναι πολύ δύσκολο κανείς να φανταστεί κάτι τέτοιο. Να, έχουμε, να έχει άμεσο αποτέλεσμα άμεση επίπτωση σε κάποιον ο οποίος ε, βλέπει ανταγωνιστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χρήσιμο περισσότερο κάτι που μπορεί ίσως να επηρεάσει κάποιον που είναι ουδέτερος ή δεν έχει εμπλακεί ιδιαίτερα να γνωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώτη φορά βλέπει ένα τέτοιο πρόγραμμα, κάτι που τον κάνει να είναι θετικά διακείμενος απέναντί του. Δεν μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του ευρωσκεπτικισμού με άλλο τρόπο παρά μόνο αυτόν νομίζω. Τώρα, μεγαλύτερο ρόλο ε, θα μπορούσε να έχει το πρόγραμμα. Στην τελευταία αξιολόγηση, ε, επί της οποίας εργαστήκαμε εγώ και η Ρίνα, ένα από τα προβλήματα που βρήκαμε ήταν ότι ήταν πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα και κάνει πολλά πράγματα, αλλά με λίγα χρήματα τελικά το νέο πρόγραμμα έχει 13% λιγότερα χρήματα για να κάνει αυτό που υπόσχεται. Το θέμα είναι λοιπόν τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Αυτό πρέπει να δούμε περισσότερο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ, Μπραντ. Ελπίζω να απαντήθηκε η ερώτησή σας για το 20% από την Κομισιόν ήδη, αλλά για να επανέλθω, επειδή ίσως δεν ήμουν αρκετά σαφής, υπάρχουν πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες για τα project που έχουν να κάνουν με τη μνήμη, ενώ μόνο το 20% του προϋπολογισμού σχετίζεται με αυτό. Το 60% λοιπόν η πλειοψηφία δηλαδή του προπολογισμού είναι για το Strand 2 ε, που έχει λιγότερες επιλογές, λιγότερες προτεραιότητες, άρα έχουμε και λιγότερες ευκαιρίε ε, για project πολιτών από μία άποψη. Ελπίζω να το διαλεύκανα αυτό και τώρα για την κυρία Γιούγκ ε, να πω ότι όντως είδαμε ότι το δυναμικό των εθνικών σημείων επαφής ήταν καλό, δεν είχαν πρόβλημα να επικοινωνήσουν, όμως είχαν λιγότερες ευκαιρίες να επικοινωνήσουν, παρόλο που υπάρχει ένα ιντρανέτ. Ε, δεν είναι ένα εργαλείο αυτό που τους βοηθάει σύμφωνα με τα όσα μας είπαν. Υπάρχει το NING που είναι ένα ειδικό εργαλείο για το Creative Europe και τους επιτρέπει να, μια, να έχουν μια καλύτερη επικοινωνία Τώρα ως προς το δυναμικό, δυνα... δυστυχώς δεν είχα χρόνο στην παρουσίασή μου να πω περισσότερα, όμως θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο τακτική επικοινωνία μεταξύ των σημείων επαφής, γιατί υπάρχει μια τυπική επαφή, αλλά δεν είναι τόσο συχνή. Υπάρχει και το newsletter, το οποίο πήγε στα διάφορα αυτά σημεία επαφής και τους γνωστοποίησε κάποια νέα. Υπάρχει και, ε, υπάρχουν και οι προθεσμίες που πολλές φορές είναι απογοητευτικές και δεν εμφανίζονται στο site, το επίσημο. Και δεν πηγαίνουν και στους ενδιαφερόμενους. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, η κυρία Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ε, ε, να ξεκαθαρίσω απλώς, επαναρχόμενοι στους στόχους του προγράμματος, ότι ο στόχος του προγράμματος ήταν ε, η ενίσχυση της κατανόησης της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το είδαμε ότι είναι αναγκαίο κυρίως με την αύξηση της, του ευρωσκεπτικισμού. Πολλοί πολίτες ε, επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν κατανοούν πώς λειτουργεί. Έτσι, ε, το πρόγραμμα στην ουσία κάτι τέτοιο προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Υπό το φως αυτών, λοιπόν, είναι ιδιαίτερα τυχαίο το γεγονός ότι έχει κοπεί τόσο πολύ η χρηματοδότηση. Κάτι άλλο που έχει να κάνει με τον ευρύτερο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αληθές ότι βάσει της νομικής βάσης ε, το Κοινοβούλιο δεν ενεπλάκει στην τακτική νομοθετική διαδικασία που είναι ατυχές δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο στην ουσία εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια αμέσως τώρα. Πρόεδρε, αυτοί που ασχολούμαστε με το πρόγραμμα αυτό είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στην Ευρώπη. Προφανώς και θα υπάρχουν λόγοι και υπάρχουν λόγοι για την απογοήτευση που αισθάνονται διάφοροι συμπολίτε μας. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά πράγματα για να είναι πιο γνωστά τα όσα κάνουμε εδώ η δουλειά μας και προφανώς και θέλουμε να συζητήσουμε με τους ε, συμπολίτες μας που ανησυχούν για αυτά τα θέματα και θα έπρεπε να ε, προωθήσουμε τέτοιο διάλογο. Και για αυτό είναι σημαντικό αυτό το πρόγραμμα, όπως και για τις ενισχύσεις στις οποίες αναφέρθηκε η κυρία Ναμάτο. Ε, το, το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαμε έρθει σε επαφή με 7 εκατομμύρια πολίτες είναι πολύ σημαντικό και σημαίνει ότι έχουμε μια, ένα μοχλό στη διάθεσή μας για να γνωστοποιήσουμε, να κάνουμε μια σωστή προώθηση όλου αυτού του έργου. Νομίζω ότι και με την βοήθεια της Κομισιόν μπορούμε να επιλύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ε, δεν θα ήθελα να επεκταθώ άλλο. Να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή και ελπίζω πραγματικά να φτάσει το πρόγραμμα σε αυτό που φιλοδοξούμε. Δηλαδή ενισχυμένο προϋπολογισμό και ενισχυμένο αποτύπωμα αν θέλετε και προϊόν. Σας ευχαριστώ και εγώ λέει Πρόεδρος για τη συζήτηση, για τις παρουσιάσεις ε, που θα μας ε, βοηθήσουν όλους που είναι πολύτιμες. Εμείς και στο σχέδιο προϋπολογισμού που μόλις ψηφίσαμε ζητήσαμε σημαντική αύξηση του σχετικού προπολογισμού και δεν θέλαμε να αποδεχθούμε την αρχική μείωση που βεβαίως σημειώθηκε αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο αρχικά προτάθηκε. Ε, εγώ νομίζω ότι η συνολική εικόνα είναι θετική. Δηλαδή πρέπει να ενισχύσουμε την συμμετοχικότητα και, την, ε, ε, και να είμαστε ανοιχτοί, όχι μόνο δηλαδή προς τους πολίτες αλλά και σε διαμένους χώρες μας, να έχουμε μια προώθηση τη συλλογική ιστορική γνώση, αλλά και της ε, ενεργού συμμετοχικότητα και της πρόσβαση, της δυνατότητας πρόσβασης ε, στην κοινή προσπάθεια για μια δημιουργία ε, μια διαφορετικής Ευρώπης. Και εδώ συμφωνώ και με συναδέλφους που δεν πρέπει απλώς να αποδεχθούμε την Ευρώπη έτσι όπως έχει, πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα και να είμαστε πρωταγωνιστές, πρωταγωνιστές σε αυτήν την Ευρώπη που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Και προς αυτό θα πρέπει να κατευθύνει τη δουλειά μας, όπως και στην ενίσχυση, την απελευθέρωση της δημιουργικότητας των πολιτών. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και την Κομισιόν. Με αυτό μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο της ημερησίας διατάξεως. Ζητώ συγγνώμη που δεν σας χαιρετώ έτσι επισήμως, αλλά έχουμε πολύ λίγο χρόνο και έχουμε και άλλο σημείο το τελευταίο της ημερησίας διατάξεως. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα δώσω λοιπόν αμέσω. μάλλον, θα περάσω στο επόμενο σημείο που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό της ε, Οικονομικής Πολιτικής. Έχουμε τον κύριο Σδρογεύσκη που βρίσκεται εδώ, που είναι ο συντάκτης. Γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο προβλέπει ε, την υλοποίηση των προτεραιοτήτων 2016 και έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την ε, αναθεώρησή τους. Θεωρούμε ότι πρέπει να επανακινήσουμε με ενεργητικότατο τρόπο σχετικά με όλες τις πολιτικές που αφορούν στην παιδεία, τη δημιουργικότητα, την εκπαίδευση, τους νέους ε, έχουμε λοιπόν κάθε συμφέρον να συμμετάσχουμε πολύ ενεργά σε αυτήν τη συζήτηση για το εξάμεινο. Τώρα, για σχέδιο γνωμοδότησης ε, αποφασίστηκε η ΕΚΟΝ και φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούν. Ε, η προθεσμία είναι 7 Σεπτεμβρίου μεθαύριο, στις 11 η ώρα, για την υποβολή τροπολογιών, γιατί πρέπει να υποβληθεί η έκθεση 11 Οκτωβρίου. Το σχέδιο έχει ήδη διαβιβαστεί από τις 13 Ιουλίου στους Σκιώδης και είχαμε ήδη επισημάνει το χρονοδιάγραμμα. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Σδρογεύσκη, θυμίζοντας ότι 26 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την ψήφο στην ε, Επιτροπή Κουλ. Του παρακαλώ, Μπόγκταν. Να 12 e, Πρόεδρε, 12 λεπτά μας μένουν. για την γνωμοδότηση αυτή και για τα διάφορα. Πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε την ευκαιρία και αυτή είναι να συζητήσει η Επιτροπή μας το εξάμεινο και να επισημάνει τρία σημεία. Καταρχάς την αξία του πολιτισμού, στη δημιουργία, απασχόλησης, οικονομικής, ε, οικονομικής δραστηριότητας και βέβαια όρων απασχόλησης για τους νέους. Ε, επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο πολιτισμός ως τομέας είναι ιδιαίτερα ε, Σημαντικό για τη δημιουργία θέσεων εργασία, Πρόκειται για ένα τομέα ο οποίο δημιουργεί περισσότερε θέσει εργασία ε, από ότι επενδύσει σε διαφορου τομεί που μπορεί να φαίνονται ε, περισσότερο σχετικοί με την αγορά ή να υπόσχονται περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, η γνωμοδότηση δεν σκοπεύω να είναι υπερβολικά μακροσκελής. Ε, θέλω να την περιορίσω σε συγκεκριμένα σημεία για να μην χαθεί και το μήνυμά της. Το κύριο αυτό μήνυμα ώστε να είναι η γνωμοδότησή μας στην Οικονομική Επιτροπή όσο το δυνατόν πιο σαφής και ευανάγνωστη. Σημειώνουμε λοιπόν ότι οι επενδύσεις τον πολιτισμό ενισχύουν τις πιθανότητες αύξησης απασχόλησης ή υποστηρίζουμε το Erasmus Plus για, μια, για την ενίσχυση απασχόληση σε όλη την Ευρώπη ή υπογραμμίζουμε τη σημασία της προαγωγής καλύτερης προαγωγής του προγράμματος και βεβαίως ο δημιουργικός τομέας, ε, ο καλλιτεχνικός τομέας, γράφουμε, ενισχύει τις πιθανότητες απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν ξέρω αν έχουμε παρατηρήσεις Μαραγκάλ, Τζούλι Βόρτ και μετά η κυρία Χιμένηθ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Gracias, Ευχαριστώ πρόεδρε. Το θέμα δεν είναι να βρούμε τα στοιχεία που θα μπορούσε να επικρίνει κανείς ε, στην έκθεση του κυρίου Σδρογεύσκη. Πάντα ε, ο κίνδυνος, αν θέλετε, είναι αυτή η τάση που έχουμε να προσθέτουμε πράγματα. Εγώ θα μπορούσα να συνοψίσω ως εκεί, ως εξής. ίσως ε, μια πιο κριτική θέση σε σχέση με την παρούσα κατάσταση του ευρωπαϊκού εξαμήνου και ιδιαίτερα προς την οικονομική πολιτική. Όπως ε, και σχετικά με τα στοιχεία που εμείς εδώ σε αυτή την Επιτροπή προσπαθούμε να υπερασπίσουμε. Έχουμε και μια υπερβολική ακαμψία του μέσου αυτού ε, ως μέσο πολιτικής ε, και ως συσχετισμό μάλλον ως πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών που καθένα έχει τη δική του φύση και δομές ε, και υπό την αυτή το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν τα κάνει αυτά. Θα πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη ελαστικότητα για να προσαρμόζεται σε αυτές τις ε, διαφορετικές προελεύσεις παραγωγικών προτύπων κτλ. Ακριβώς υπό την έννοια αυτή η επένδυση στην παιδεία και στον πολιτισμό προσφέρει διάφορες θαυμάσιες λύσεις εάν ποτέ η Κομισιόν θα ήθελε να εντάξει στο πλαίσιο αυτό τα κριτήρια και τις στρατηγικές που υπερασπιζόμαστε. Και στις τροπολογίες μας ακριβώς προσπαθούμε να υπογραμμίσουμε κάποιες από αυτές τις δυνατότητες. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να μην σημειώνουμε ότι με τις πολιτικές λιτότητες που το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αν θέλετε, εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή, έχουμε καταφέρει στις χώρες που πιο απαραίτητες θα ήταν αυτές οι πολιτικές προκειμένου να βγούνε από την κρίση, εκεί ακριβώς σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες περικοπές στους προϋπολογισμούς παιδείας και πολιτισμού, το οποίο είναι σκανδαλώδης αντίφαση. Θα πρέπει λοιπόν να αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Κομισιόν υπό την έννοια αυτή, ότι δηλαδή ο τομέας της παιδείας και του πολιτισμού Διακόπτη πρόεδρος, συντομεύεται. Έλεγα λοιπόν για να ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλοι τομείς που έχουμε ξεχάσει είναι πολύ γόνιμο πεδίο για την έξοδο των χωρών από την κρίση. Και βεβαίως ο ρόλος της μετανάστευσης και των δυνατοτήτων που δίδει εάν αναπτυχθούν πολιτικές παιδείας που να συνάδουν τους ανάγκες των χωρών. Ελπίζω λοιπόν ε, οι προτάσεις μας και ε, οι τροπολογίες να βρουν το χώρο που χρειάζονται. Σας ευχαριστώ, η ε, κυρία Ward. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο και φαίνεται ότι η ζημιά που έχει κάνει η λιτότητα στους νέους ειδικά είναι κάτι με το οποίο όλοι συμφωνούμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δημιουργήσουμε και να προωθήσουμε δουλειές υψηλής ποιότητας ασφαλής θέσεις εργασίας σύμφωνα με την ατζέντα του ILO. Οι πολιτικές για τις οποίες μιλώ θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της επισφαλούς εργασίας μέσα από προγράμματα ε, στάζ, μέσα από ε, προγράμματα που θα αντιμετωπίσουν, ας πούμε, τις περικοπές στο δημόσιο τομέα. Επίσης, η κοινωνική εταιρικότητα και επιχειρηματικότητα είναι ένας τομέας που υπόσχεται πολλά, γιατί δένει τις κοινότητες μεταξύ τους, ε, ε, οδηγεί στην κοινωνική ενσωμάτωση και την αντιμετώπιση της ανέχειας. Έχουμε το fair trade, ε, τις κοινωνικές επιχειρήσεις με εναλλακτικά μοντέλα, εταιριών και συνεταιρισμών. Επίσης, η κινητικότητα σε άτυπα και τυποποιημένα πλαίσια, ειδικότερα των νέων που δεν προέρχονται από, πλεονεκτικές, ε, από πλεονεκτικό υπόβαθρο. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν τους νέους, ε, τους ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν στις αντίστοιχες βιομηχανίες. Ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο μας, λέει η Πρόεδρος, ε, ο συνάδελφος, η Μπαρμπάτ και μετά η κυρία Νίκο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σχετικά με το σχέδιο της ε, γνωμοδότησης, οι προοπτικές ανάπτυξης ε, αυτή τη στιγμή είναι αδύναμες και βρίσκονται σε ένα πλαίσιο αμφίβολης εξέλιξης οικονομικής έχουμε σημαντικά τμήματα του πληθυσμού, όπως ιδιαίτερα οι νέοι, που υποφέρουν ε, ιδιαίτερα από την κρίση αυτή και ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σδρογεύσκη ως εισηγητή της Επιτροπής ε, Πολιτισμού γιατί γνωρίζει αυτές τις ε, προκλήσεις και αυτά τα προβλήματα και γνωρίζει ότι πρέπει να επιληθούν αυτά να αντιμετωπιστούν το συνημότερο δυνατόν προκειμένου να είναι πιο ανταγωνιστικά στην εξωτερική αγορά τα κράτη-μέλη, χρειάζεται να επενδύσουμε με ευφυή τρόπο στην ε, παιδεία και τον πολιτισμό, αλλά και στους ε, πολίτες, στους Ευρωπαίους πολίτες και στην κοινωνία των πολιτών. Και στις τροπολογίες μου ιδιαίτερα τονίζω το ρόλο που πρέπει να ρεματίσει η επιστήμη ε, και η θρησκεία σε αυτό το πλαίσιο. Και χρειάζομαστε τον ορίζοντα του 2020, χρειαζόμαστε η επιστημονική κοινότητα να συνεισφέρει σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία, ώστε να υπογραμμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πορείας ε, συνεργασίας διεθνώς και ανάπτυξης. Πολύ συχνά ξεχνούμε τα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη σημασία τους για τους ε, πολίτες, για τους ε, σπουδαστές και τη συνεισφορά τους στην οικονομία της Ευρώπης, όπως και για την σημασία που έχει η κοινωνία των πολιτών και ενσωμάτωσή της στο ραϊκό σύστημα. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Στρέσκη για τη δουλειά του. Με τη γνωμοδότηση αυτή, όπου διαβάζω πράγματα ενδιαφέροντα με τα οποία συμφωνώ ε, παραδείγματι διαβάζουμε ότι έχει μειωθεί σε σχέση με πέρσι το ποστό ανεργίας των νέων. Παραμένει ωστόσο ανησυχητικό το φαινόμενο και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της απασχόλησης, γιατί η ποιοτική απασχόληση μπορεί να επιτρέψει την επίλυση των προβλημάτων της ενεργείας. Επίσης έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπε και ο εισηγητής για τον προσανατολισμό προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει βεβαίως να δούμε τις μεταρρυθμίσεις και ε, εν των αναγκών των, των επιχειρήσεων, αλλά και εν ώψη των κοινωνικών αναγκών. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν υπάρχουν ε, στάδια Φερρυπίν ενδιάμεσα που θα επέτρεπαν στον νέο να εξασφαλίζει και την ε, καλή θέση εργασίας και την ε, κοινωνική προστασία. Γενικά πρέπει να έχουμε ένα καλό σύστημα κατάρτισης, πρακτικής, εκπαίδευσης, αλλά και κάθε άλλη μορφή κατάρτισης, εκπαίδευσης που μπορεί να αποτελεί ε, χρήσιμο εργαλείο και που μπορεί να προβάλλει η ε, Επιτροπή μας. Επίσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020 θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους που βρισκόνται σε δύσκολη κατάσταση. Μητέρες, ε, ιδιαίτερα μετά την ε, περίοδο της άδειας μετρότητας, να επανεντάσσονται στον στο χώρο της εργασίας. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα για να επιτύχει το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Και παρακαλώ να μας κάνετε τα σχόλιά σας. Και εσείς ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα σχόλια. Μερικές ε, παρατηρήσεις για τις συζητήσεις που έγιναν. Καταρχάς πιστεύω ότι η στρατηγική είναι μια στρατηγική η οποία επιδιώκει ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την απασχόληση. Άλλωστε το έχει υπογραμμίσει και ο πρόεδρος Γιούγκερ στις, κατα... στις γραμμές. Όχι μόνο δηλαδή την πτυχή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά και τις κοινωνικές πτυχές θέλει να υπογραμμίσει η Επιτροπή. Και έτσι συνδυάζουμε την απασχόληση, στα κοινωνικά αισθήματα, την ανάπτυξη. Και βέβαια αυτό ήταν πάντα και το πνεύμα το οποίο καθοδηγεί τις ε, επενδύσεις και θα υπάρχει η εξυγίανση δημοσιονομική αλλά αυτή δεν θα γίνεται βεβαίως κατά τρόπο τυφλό και γενικό, ε, σαρωτικό. Θα γίνεται η δημοσιονομική εξυγίανση κατά τρόπο να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη, το μέλλον της οικονομίας. Και βεβαίως έτσι έγιναν δεκτές και οι προτάσεις ε, σε επίπεδο επιτροπή και σε επίπεδο Συμβουλίου. Ε, μεγάλο ρόλο θα δερματίσει αυτά η εκπαίδευση, ο πολιτισμός που αναφέρατε και εσείς, η κινητικότητα, η διαφάνεια μια σειρά συστάσεων προς τα κράτη-μέλη, υπογραμμίζει ιδιαίτερα τις κοινωνικές, τα κοινωνικά ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες ε, ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, νέων ε, που χρειάζεται να μπουν ε, μέσα στο σύστημα του εργασιακό, Ρωμά, ατόμων που προέρχονται από τη μετανάστευση. και έτσι χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως σημειώνουμε που θα εξασφαλίσουν και ισορροπία στην ανάπτυξη, αλλά και συνδυασμό ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτά είναι τα διάφορα σημεία λοιπόν που ε, επισημαίνει και το σχέδιο γνωμοδότησής σας. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την αντιμετώπιση του φαινομένου της εγκατάλειψης, πρώιμης εγκατάλειψης του σχολείου, τι μπορεί να κάνει ο διδάσκον, παραδείγμα, τι πώς μπορεί να βοηθήσει, τι συνεργασία μπορεί να υπάρχει μεταξύ σχολείου και επαγγελματικών ε, διεξόδων, λύσεις δηλαδή και ιδέες που έχουν να κάνουν και με την ανάπτυξη αλλά και με την κοινωνική προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πιστεύουμε ότι ε, παρουσιάζει μια αρκετά ισορροπημένη εικόνα ως πρόταση από πλευράς μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you so much. And now uh, the... Ευχαριστώ πολύ και τώρα δίνω το, δίνω το λόγο στον εισηγητή για να ολοκληρώσει. Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ πολύ όλους ε, όσοι παρουσίασαν ε, κάποιες παρατηρήσεις. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Τώρα περιμένω την κατάθεση των τροπολογιών. Θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη όλες ε, τις παρατηρήσεις για να γίνουμε όλο και πιο, όσο πιο γρήγορη γίνεται, πιο ξεκάθαρη γίνεται, συγγνώμη. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στην Καταρχά την πρώτη, στην επόμενη συνεδρίαση 26 ε, Σεπτεμβρίου 3 ε, με 6.30 να ευχαριστήσω όλους έχουμε ακόμα εδώ τους Γερμινείς και επομένως θα μπορούμε να περάσουμε τώρα στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών γιατί χρειαζο... έχουμε κάποια σημαντικά πράγματα και θα έχουμε κάποιο χρόνο τώρα για να τα δούμε με ησυχία. Παρακαλώ τους υπόλοιπους συναδέλφους να αποχωρήσουν τώρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τους συντονιστές.